Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινώ τη συνεδρίαση. Σα εύχομαι το καλώ όρισε Πρώτα απ' όλα στους στον Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ράινερ Βίλαντ, υπεύθυνο για τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένα θερμό καλώ όρισε και στον Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριο Κλάου Βέλε. Και πριν να περάσουμε στο μόνο θέμα της ημερήσιας μας διάταξης, την ε, συζήτηση δηλαδή για τον πιθανό προϋπολογισμό για το 2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σας καλέσω να εγκρίνουμε, εάν δεν έχετε αντίρρηση, το αίτημα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που έχει ένα πρόβλημα σε σχέση με το οργανόγραμμά του, κατεπήγον μάλιστα, και αν δεν έχετε αντίρρηση θα προσθέσουμε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ή παρατηρήσεις από πλευρά σα, θα συζητήσουμε και αυτό το σημείο. Και έτσι, περνάμε στην ε, καρδιά της σημερινής μας συνεδρίασης. Το προσχέδιο σχεδίου του προπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το 2017. Ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου Ντάβιτ Μαρία Σασόλη, ε, επίση υπεύθυνο για τον προπολογισμό αντιπρόεδρο, ε, υπεύθυνο για τον προπολογισμό προέδρου, ο οποίος έχει να παρουσιάσει ένα σχέδιο έκθεση στο πλαίσιο του τετάρτου πακέτου τετάρτης θέσμης μέτρων για τα σιδηροδρομικά. Εάν δεν έχετε αντίρρηση, ακούμε τον εισηγητή πρώτα, τον κύριο και μετά τον αντιπρόεδρο Ράινερ Βίλαντ. Παρουσίαση στη συνέχεια από το Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για περίπου 20 λεπτά όλα αυτά και θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και αποκρίσεις για να διπτώσουμε μετά τα συμπεράσματα. Ο κύριος Ταγάν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συνέβαλαν στην έκθεση αυτή. Σκιώδεις ηγητές, το Γενικό Γραμματέα κύριο Βέλε, τον πρόεδρο της Επιτροπής μας, πολλούς συναδέλφους και βέβαια το προσωπικό μας που εργάστηκε στο σχέδιο αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά. Οφείλω να ομολογήσω ότι πίστευα πως η έκθεση αυτή θα ήταν ευχερής, αλλά Διαψεύστηκα. Περίμενα ότι θα ήταν μια από τις συνηθισμένες αντιπαραθέσεις όπου οι ε, πολιτικοί, οι ευρωβουλευτές επιδιώκουν να επιδείξουν στους ε, ψηφοφόρους τους ότι είναι πολύ επιτυχής στην ε, αναζήτηση μικρότερου κόστους. Και από την άλλη θα είχαμε τη γραμματεία και τους αντιπροέδρους που θα προσπαθούσαν να αποδείξουν πως ένα καλώς νοούμενο κοινοβούλιο μπορεί να εργάζεται μόνο εάν έχει την κατάλληλη χρηματοδότηση. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν με τις τροπολογίες δεν έχουν ακόμη καλυφθεί στην έκθεση. Και βεβαίως, εγώ θέλω πολύ περισσότερη διαφάνεια, όχι μόνο για την κοινή γνώμη, αλλά διαφάνεια και μέσα στο Κοινοβούλιο. Χάρη στο Γενικό Γραμματέα και την αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα κυρία Ρατή, όπου συζητήσαμε σήμερα το πρωί τα θέματα της ασφάλειας, δε ευαίσθητα αυτά τα θέματα της ασφάλειας, μπόρεσα να ενημερωθώ και να γίνω σοφότερος με βάση ε, δεδομένα για το τι χρειάζεται να γίνει. Μακάρι να ήμουν σαν τον Ελμάρ Μπροκ, παλιόψημένο πολιτικό που γνωρίζει καλά τον τρόπο λήψης των αποφάσεων από το 1999 και μετά αλλά δεν είμαι τόσο παλιός και ίσως κάποιες από τις διατυπώσεις χρειάζονται βελτίωση εδώ. Η γενική προσέγγιση της αναλογικότητας ως θέμα και για το ποσό που αφορά τα νέα μέτρα ασφαλείας μέσα στο γενικό προϋπολογισμό είναι και ο λόγος για τον οποίο θέλω ιδιαίτερα να ε, επιμείνω ότι χρειαζόμαστε περισσότερη πληροφορία όχι μόνο εγώ αλλά όλοι οι συνάδελφοι της Επιτροπής. Περισσότερη ενημέρωση λοιπόν και πληροφορίες και για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε στους συναδέλφους μας από τις διάφορες πολιτικές ομάδες τις προτάσεις. Γιατί είναι ενδιαφέρον αρκετά το πώς κάθε μέλος σε αυτή τη τελική διαδικασία του δημοσιονομική εστιάζεται όλο και περισσότερο ο καθής, όπως έλεγα, σε μια πιο περιορισμένη πτυχή της καθημερινής μας ζωής. Και αν δεν είμαστε θέσει να εξηγήσουμε την πραγματικότητα, δεν είναι εύκολο να εξασφαλίσουμε και την υποστήριξη μιας πολιτικής ομάδας. Συμφωνώ με την προσέγγιση του Γενικού Γραμματέα. Τον τίτλο άλλωστε το αναφέρουμε ενίσχυση της ε, εντολής των βουλευτών. Βεβαίως αυτό είναι αυτονόητο, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να κοιτάξουμε τι σημαίνει η ενίσχυση της ε, ε, εντολή των βουλευτών όταν πρόκειται για τις εκλογικές περιφέρειες, δυνατότητα για κάλυψη εξόδων γραφείων και το καθεξής. Πάντα ήταν η στεγαστική πολιτική ένα πρόβλημα ανεπίλητο για μένα, γόρτιο θεσμό ω γι' αυτό μένω σε νοικιασμένο διαμέρισμα και δεν έχω αγοράσει δεν έχω χτίσει σπίτι. Αλλά είναι και αυτό ένα από τα ζητήματα που θα μα απασχολήσουν στη δημοσιονομική διαδικασία και ιδιαίτερα θέλω να αναφέρω την προβλεπόμενη ανακαίνιση του κτηρίου Paul Henry Spack. PHS. Θα ήταν καλό να γνωρίζουμε λοιπόν τι ανάγκες υπάρχουν, τι αναλύσεις και αξιολογήσεις ή εκτιμήσεις μπορούν να γίνουν για να λάβουμε τις σχετικές αποφάσεις με τα γνώσεις λόγου. Η υπηρεσία των οδηγών επίσης. Και πάλι ευχαριστώ τους Κιώδης, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν με πολύ ενδιαφέρον. Ήρθαν ακόμα και πολύ πρωινές ώρες να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Δεν θα έλεγα ότι το καταλάβαμε πώς ακριβώς παρουσιάστηκε. Γι' αυτό στην έκθεση, παρά τις προειδοποίησεις που γίνονται από τους πιο σοφούς ε, βουλευτές, δεν θα έπρεπε να το προσπεράσουμε, θα έπρεπε να μας δοθεί ο χρόνος να το συζητήσουμε δεξιωδικά. Το τελευταίο τώρα είναι η συνεργασία ανάμεσα το Κοινοβούλιο και τις διάφορες επιτροπές, δηλαδή την ε, Επιτροπή των Περιφερειών και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Εδώ πιστεύουμε ότι πρέπει να στηρίξουμε την ε, συνεργασία που μπορεί να υπάρχει και τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει σε αυτούς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ερωτήσεις βάζουμε. Εγώ προσωπικά έτσι μαθαίνω. Κάνω ερωτήσεις. Οι απαντήσεις που πήραμε μέχρι τώρα ήταν καλές και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Βέβαια είναι ίσως εύκολο όταν είναι χαζές οι ερωτήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στρατηγική εγώ ακολούθησα για την εκπόνηση της εκθεσής μου. Εδώ θα ολοκληρώσω, δεν χρειάζεται να πω εγώ περισσότερα, καλύτερα να μιλήσουν οι διάφοροι ομιλητές, δηλαδή και από το Προεδρείο και τη Γραμματεία, αλλά και οι συνάδελφοι εδώ στην Επιτροπή αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Σιγητά που μοιραστήκατε μαζί μας τις πολύ καλές ερωτήσεις σας. Ο πρόεδρος διπρόεδρος Βίλαμε έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε και ευχαριστώ αγαπητέ κύριε Τάραντ για την ε, εισαγωγή στο θέμα. Εγώ από πλευράς μου θα ήθελα να πω ότι μου φαίνεται ιδιαίτερα θετικό το ότι δεν βλέπω κατά αποκοπήν ποσά και ε, αυθαίρετες ε, αριθμητικές παραστάσεις μέσα στην έκθεση. Βλέπουμε σε ορισμένα σημεία δηλαδή στο σημείο 13 παραδείγματι ότι εκφράζονται και θετικά σχόλια και θα ήθελα ιδιαίτερα να χαιρετήσω το γεγονός ότι και εσείς στον τομέα των, ε, της ε, μηχανογράφησης και της εξυπηρέτησης με ηλεκτρονικούς υπολογιστές το 2017 μας λέτε ότι είναι ένα κομμάτι της δουλειάς μας που δεν μπορούμε να παραμελήσουμε. Τώρα το αν θα πρέπει να καταργηθούν οι συσκευές τηλετύπου, τα φαξ, μπορούμε να το συζητήσουμε. Ίσως κάποιοι από τους πιο παλαιούς βουλευτές να αμυνθούν εναντί αυτής της προτάσεως. Εγώ από τη δική μου τη σκοπιά ήθελα να κάνω κάποια σχόλια περιοριζόμενος όμως σε συγκεκριμένους τομείς και ίσως θα τονίσω μόνο τα πιο σημαντικά σημεία, αυτά που χρειάζονται, ε, χρειάζεται να εξεταστούν ως προτεραιότητες. Το 2016 θα χαρακτηριστεί νομίζω ως το έτος το οποίο μας απασχόλησαν περισσότερο από κάθε άλλη φορά ζητήματα ασφάλειας. Χρειάζεται να καλύψουμε χαμένο έδαφος. Είδαμε στα τέλη του προηγούμενου έτους της, την προσαρμογή στην ε, είσοδο από την πλευρά της πλατείας Λουξεμβούργου, στη συνέχεια από την ε, πλευρά της Οδουβίρτς Θα συνεχιστούν αυτά. Θα δούμε μέτρα τα οποία ίσως να μην επηρεάσουν ιδιαίτερα την καθημερινή ζωή των βουλευτών, όσο η ε, αλλαγή στο σύστημα των εισόδων, αλλά πάντων θα είναι Παντώ θα είναι και άλλα μέτρα αντίστοιχα για την ενίσχυση της ασφάλειας σε κάθε σημείο τη αλυσίδα για να ενισχυθούν και οι πιο δύναμοι ακόμη κρίκοι της αλυσίδα της ασφάλειας. Και θα πρέπει να κοιτάξουμε και τις εισόδους με το απλό τζάμι, όπου ίσως χρειάζονται ενίσχυση εν πάση περιπτώσει θα μας απασχολήσουν περαιτέρω και για το 2017 και στη συνέχεια ίσως τα ζητήματα τα ακτηριακά. το τι θα κάνουμε με το προσωπικό ασφαλείας, το αν θα έχουμε μέσα στο Κοινοβούλιο ένοπλους φρουρούς, παραμένει εκκρεμές. Παραμένει επίσης το εάν θα έχουμε διαφορετικές βαθμίδες ασφαλείας ή επιφυλακής καλύτερα και σε περίπτωση αυξημένων συνθήκων ασφαλείας εάν θα πρέπει να έχουμε αστυνομικές αρχές ή και στρατιωτικές δυνάμεις. Αυτά είναι ζητήματα όχι μόνο πολιτικά αλλά και οικονομικά έχουν οικονομικό αντίκτυπο. Το Κοινοβούλιο πάντως θα πρέπει να βρει τα σχετικά κονδύλια. Ε, τροποποιήσεις επίσης στα κτίρια τα οποία θα μας απασχολήσουν πιστεύω στην επόμενη πενταετία και που θα σημάνουν μεγαλύτερες επενδύσεις ή πάντως κόστος και τα, θα απαιτήσουν τα απαραίτητα τα σχετικά κονδύλια. Άρα λοιπόν οι επενδύσεις ε, οι οποίες θα καλύψουν αυτές τις ανάγκες στην ασφάλεια. Θα πρέπει να δούμε αν θα υπολογιστούν μέσα στον προπολογισμό, αν θα βγουν κατά κάποιο τρόπο από αυτόν. Και μέσα σε αυτό έρχεται και η πολιτική για τα κτίρια, γιατί δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η πολιτική για τα κτίρια χωρίς να συνδεθεί με την πολιτική για την ασφάλεια. Και μεγάλη σημασία εδώ θα έχει Μεγάλη σημασία λοιπόν θα έχει το πώς θα συνεχίσουμε από εδώ και πέρα. Το 2017 δεν θα έχουμε μεγάλα κονδύλια και είναι απαραίτητο να γίνεται εγκαίρος ο προϋπολογισμός και ο προγραμματισμός των δαπανών. Εγώ θέλω να υποστηρίξω να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο αυτό το ζήτημα, να το συζητήσουμε και να το μελετήσουμε ακόμη περισσότερο και βέβαια μεγάλη σημασία έχει το πότε ξεκινάμε τις πρώτες μεγάλες εργασίες εξυγίανσης των κτηρίων, το PHS μετά το ASP θα χρειαστεί να προχωρήσουμε μέσα από τη διαδικασία αυτή της εξυγένσης και ασφαλώς για τα 2019-2024 θα μας απασχολήσουν αυτές οι εργασίες. Ίσως δε η περίοδος ε, γύρω από τις εκλογές να ε, μας φανεί χρήσιμη για να κάνουμε τις σχετικές προσαρμογές. Και ίσως θα καλό και να μας απασχολήσει το τι θέλουμε να κάνουμε τελικά με τα κτίρια αυτά. Θέλουμε ως το δυνατόν ε, περιορισμένη ανακαίνιση, παύλα εξυγίανση. Πράγμα το οποίο εγώ από προσωπική πείρα ξέρω ότι δεν έρχεται και τόσο εύκολα. Εγώ έχω γραφείο στον 11ο όροφο και είδα μέσα ποντικό. Δεν είναι εύκολο να φτάσει στον 11ο όροφο ένα ποντικό από μόνο του, άρα κάτι άλλο κρύβεται πίσω από αυτό. Και υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έκαναν λόγο για αρουραίο μέσα στο κτίριο. κτίριο είναι ένα κτίριο που έχει κάποια χρόνια πίσω του και δεν έχει σχεδιαστεί για τη χρήση στην οποία έχει έρθει τώρα. Έχουμε επίσης γύρω από το κτίριο του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο εγκαταστάσει, οι οποίε έχουν ηλικία 20, 25, ακόμα και 30 ετών. Ή έχουμε ε, εξοπλίσει ε, εκ των υστέρων φυσικά λόγω της εξέλιξης τεχνολογίας με ίντερνετ τα κτίρια μέσα ε, με καλώδια τα οποία φτάνουν και τα 100 χιλιόμετρα ακόμα έγιναν εκ των υστέρων όλα αυτά. Λοιπόν, χρειάζεται κάποια εξυγίανση και πρέπει να δούμε σε ποιον θα την, θα την αναθέσουμε. Έχουμε να κάνουμε με ε, παράθυρα που πρέπει να αλλάξουν, κάποιες πόρτες που δεν κλείνουν ή τρίζουν. Ε, θα περιοριστούμε μόνο σε μια διορθωτική ε, παρέμβαση ή θα θελήσουμε να κάνουμε μια αλλαγή η οποία θα μας φέρει σε ένα ακόμη πιο προχωρημένο στάδιο για ένα ε, παθητικό ενεργειακά κτίριο, ένα κτίριο το οποίο θα καλύπτει και όλες τις ανάγκες σε ασφάλεια. Ή μήπω θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το Caprice de Dieu, το περίφημο αυτό θόλο που έχει το, το κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες που ε, έχει όγκο μερικών εκατοντάδων κυβικών μέτρων και δεν αξιοποιείται. Μήπως θα έπρεπε να κοιτάξουμε να το αξιοποιήσουμε αυτό. Άλλε αίθουσε συνεδριάσεων ίσω χρειαστούμε. Δεν μπορούμε να έχουμε αίθουσε συνεδριάσεων με μόνο δύο ή τρει γλωσσε δυνατοτητα δυνατότητα κάλυψης δηλαδή δύο-τριών γλωσσών. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να σα απασχολήσουν το 2016. Ξεκινάμε τη δουλειά αυτή φέτο. Έχετε δίκιο. Αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τον προπολογισμό του 19 ήδη. Με αυτά που θα μα απασχολήσουν. Και επίση, η υπηρεσία των οδηγών, που πολύ σωστά επισημάνατε. Τα λέω ακόμα και αν μεταδίδομαι από το διαδίκτυο δεν έχουμε τη δυνατότητα εδώ στο Βελγίο και με δεδομένες ε, τις δυνατότητες εξυπηρέτησης από ιδιωτικές επιχειρήσεις εδώ στο Βέλγιο να αναθέσουμε την κάλυψη των αναγκών μας σε αυτοκίνητα με οδηγό όπως θα μπορούσαμε φερρυπίν να το πράξουμε στο Βερολίνο, στη Γερμανία. Υπάρχει περιορισμένη προσφορά αυτής της υπηρεσίας, μερικές δεκάδες χιλιόμετρα το χρόνο μόνο, που θα μπορούσαμε να ε, εξασφαλίσουμε ως ε, υπηρεσία με διαγωνισμό σε εξωτερική ιδιωτική δηλαδή εταιρεία. Αν κάποια μέρα λοιπόν έρθει ε, ο πρόεδρος της γερμανικής δημοκρατίας να ε, κάνει μία επίσκεψη, μία όμορφη μέρα ανοιξιάτη και αποφασίσει να βγει το Σάββατο μία βόλτα και χρειάζεται να το συνοδεύσουν κάποιοι, δεν θα έχουμε αρκετά αυτοκίνητα ή θα πρέπει να παραγγείλουμε ταξί, γιατί εταιρείε με οδηγό δεν υπάρχουν αρκετέ. Ή αλλιώ θα πρέπει να κοιτάξουμε άλλε λύσει ή να μιλήσουμε για εσωτερική υπηρεσία οδηγών. Είναι κάτι που μας απασχόλησε και πριν από 5 ή 6 χρόνια με την κυρία Λούλινγκ, την κυρία Ροτ Μπέρεντ. Πήγαμε, είδαμε και τι δυνατότητε που προσφέρει το Βερολίνο ω πόλη και διαπιστώσαμε ότι εδώ στις Βρυξέλλε θα είχαμε τη δυνατότητα για τέτοιου είδου διαγωνισμούς με ανάθεση τη σχετική ε, σύμβασης για την κάλυψη των αναγκών μας σε αυτοκίνητα με οδηγό εδώ στις Βρυξέλλε. Αυτό είναι λοιπόν το ένα, το σημείο 14. που ξεκινήσαμε λιγότερο φιλόδοξα αλλά καταφέραμε αρκετά πιστεύω με την κυρία Ρατή και στο σημείο 12 όπου θα ήθελα να δω μια αιτιολογία τουλάχιστον στις ε, τοποθετήσεις γιατί έχω την αίσθηση, την αίσθηση ότι έχουν γίνει χειρότερα τα πράγματα. Έχουν χειροτερέψει. Ίσως βέβαια αυτό αποδίδεται και στο γεγονός ότι τους τελευταίους τέσσερις μήνες έχουμε αυτούς τους περιορισμούς στην είσοδο μας, κατά την είσοδο μας στα κτίρια. Και πρόεδρε, στο συγγνώμη γιατί ξέχασα δύο πράγματα να αναφέρω. Πρώτον, δεν πιστεύω ότι η να αποζημίωση μπορεί να αποτελέσει έναν τρόπο εξοικονόμησης κονδυλίων μάλλον η αλλαγή από το σύστημα της καταποκοπήν ε, αποζημίωσης θα μπορούσε να σημάνει πραγματικά εξοικονόμηση πόρων για το Κοινοβούλιο. Έτσι θα χρειαζόμασταν ένα μεγάλο αριθμό υπαλλήλων που θα επαλήθευαν τις δαπάνες των βουλευτών. Άρα έχει κάποιο νόημα η καταποκοπή αποζημίωση. Εσείς κύριε Τάραντ, ίσω θέλετε να κοιτάξετε ένα έγγραφο το οποίο έχω συμπηλήσει στα γερμανικά Δυστυχώ, δεν είχα τη δυνατότητα να το μεταφράσω, αλλά έχουμε το Συνταγματικό Δικαστήριο της Καλσρούης της Γερμανίας, το οποίο με μια πρόσφατη αποφασή του ε, όχι μόνο ε, χαρακτήρισε νομικά ε, νομοθετικά δηλαδή παραδεκτεί αυτή τη μέθοδο της καταποκοπήν αποζημίωσης για βουλευτές, αλλά δίνει και οικονομικές ερμηνείες και επιχειρήματα. Και το δεύτερο που ήθελα να, να προσθέσω έχει να κάνει με τα νούμερα που έχουμε στη θέση μας, τα αριθμητικά στοιχεία για το MEP ranking, για την ταξινόμηση δηλαδή της δραστηριότητας των βουλευτών. Εγώ είμαι πεπισμένος πολέμιος της ποσοτικής προσμέτρησης των επιδόσεων των βουλευτών. Έχουμε βουλευτές οι οποίοι μπορεί να έχουν καταγράψει και 900 τοποθετήσεις, εκατοντάδες τροπολογίες προφορικές ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες χίδιν θα έλεγα παράγονται, πολλές φορές μάλιστα. Χωρίς ε, καν να επιδιώκουν μια πραγματική απάντηση, αλλά απλώς την ε, συμπλήρωση ποσοστών και στατιστικών που θα έδιναν μια καλή εικόνα για τον βουλευτή. Νομίζω λοιπόν και πρέπει να το ζητήσουμε, να κοιτάξουμε πραγματικά την ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου, το, η οποία δείχνει πάρα πολύ ωραία ποιες είναι οι δραστηριότητές μας. Δεν είναι απαραίτητο να κοιτάξουμε το κάθε, ε, στο κάθε κεφάλαιο τα ποσά, τα νούμερα δηλαδή, τα αριθμητικά στοιχεία, τα οποία ε, δείχνουν ε, πόσες τοποθετήσεις, ομιλίες και περωτήσεις έχει κάνει ο καθένας. Αν κοιτάξτε τη δική μου την ιστοσελίδα, παραδείγματι, αν ήταν στο Βίλαντ, εγώ όταν προεδρεύω στο κοινοβούλιο τι είμαι, κάνω ομιλία ή δεν κάνω, δίνω το λόγο στον έναν και στον άλλο. Αυτή δεν είναι η δουλειά μου ως πρόεδρου, ως προεδρεύοντας τη συνεδρίαση. Θα μετρήσει λοιπόν αυτό. Κοιτάξτε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Διαφορετικά θα μπορούμε να έχουμε ε, και όταν ε, θέλουμε να έχουμε το web stream, πρέπει να έχουμε και το προσωπικό, το σχετικό, τον ε, ηχολήπτη, τον ε, κάμεραμαν και ούτω καθεξής. Ε, πρέπει λοιπόν να έχουμε και την ευθύνη να πούμε ότι να, ο αντιπρόεδρος που προεδρεύει δεν θα ψηφίσει. Εκείνος ο οποίος ασθενεί ή ε, μια βουλευτής γυναίκα η οποία είναι τιμόγενη δεν θα συμμετάσχει στην ψηφοφορία. Όλα αυτά πρέπει να τα πούμε ξεκάθαρα και μπορούμε να πούμε απλούστατα σβήνουμε τα στοιχεία για να μην χρειάζεται να τα ψάχνουμε όλα αυτά ένα-ένα και να τα επαληθεύουμε. Απλώς τα σβήνουμε, σβήνουμε την αναφορά τέτοιων αριθμητικών στοιχείων από την ιστοσελίδα. Και σε τόσο όποιος θέλει να του καταγράφουμε τα... Ε, να καταγράφονται μάλλον οι παρεμβάσεις του, ας κάτσει να τις μετρήσει μόνος του. Δεν θα τα βάλω εγώ μέσα στην ιστοσελίδα, να έχω κάποιον άνθρωπο να τα μετράει. Κύριε Τάραντ, το να πούμε ότι διευρύνουμε και εμβαθύνουμε στην ε, καταμέτρηση αυτή την αριθμητική, είναι παράνοια για ένα κοινοβούλιο. Βεβαίω εσεί ε, μπορεί να το επιδιώκετε για λόγου διαφάνεια, αλλά είναι χήμερα, είναι ένα που κάμισο αδιανό. Είναι σαν να προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι το άπιαστο. Είναι worst governance. Κάκιστη, χείριστη διακυβέρνηση και όχι άριστη διακυβέρνηση. Και γι' αυτό, εάν είχαμε και τη δυνατότητα μάλιστα να κάνουμε μια εξομοίωση των αποτελεσματικών ε, της αποτελεσματικότητας των ε, πράξεων των βουλευτών. 17.000 ήταν οι επεξηγήσεις ψήφου μέσα σε μια πενταετία για όλους τους βουλευτές. 17.000. Εάν αυτέ λοιπόν και ιδιαίτερα οι υπερωτήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν οι υπερωτοί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, περιοριστούν αριθμητικά, ίσω θα μπορούσαμε να έχουμε και το δικαίωμα να διεκδικήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την απάντηση σε αυτέ. Αν έχουμε πενταψήφιε ε, Και 24 ώρε την εβδομάδα, την ημέρα να δουλεύουν οι υπάλληλοι τη Επιτροπή, δεν προλαβαίνουν να βγάλουν απαντήσει. Δεν είναι καλή δουλειά αυτό. Πρέπει να φύγουμε λοιπόν, να ξεφύγουμε από την ποσοτική προσέγγιση. Ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό να εκτιμήσει κανείς την απόδοση, τις επιδόσεις δηλαδή. Πραγματικά δεν πρέπει να μπερδεύουμε τους δείκτες με την πραγματική επίδοση. Ο Γενικός Γραμματέας τώρα. Κύριε Γενική Γραμματέα, θέλετε να μας παρουσιάσετε τις κύριες γραμμές του σχεδίου προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι όπως τον προετοιμάσατε για το 2017. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα σύντομα να σας πενθυμίσω το χρονοδιάγραμμα, προσχέδιο δηλαδή για τον προϋπολογισμό, το οποίο κατατέθηκε σε εντατική διαβούλευση την 1η Φεβρουαρίου στο Προεδρείο. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με την Επιτροπή των Προϋπολογισμών. Στη συνέχεια θα επανέλθει για να ασχοληθεί στις 7 Μαρτίου πλέον το Προεδρείο με την πρόταση αυτή όπως θα έχει προχωρήσει μέσα από τη διαβούλευση και φανταζόμαστε ότι θα γίνει και μια επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ Προεδρείου και Επιτροπής των ε, Προϋπολογισμών και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία με την ψηφοφορία στην Ολομέλεια στις 14 Απριλίου. Ξέρετε ότι δύο δεκαετίες και περισσότερο ακόμη έχει παραδοσιακά τη διεκδίκηση το Κοινοβούλιο, 20% των διοικητικών του δαπανών 20% ε, των διοικητικών δαπανών του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού να, να ε, προορίζονται στις δικές του ανάγκες. Τώρα έχουμε φτάσει όχι στο 20% αλλά στο 19,26% των ευρωπαϊκών διοικητικών δαπανών, το χαμηλότερο δεύτερο σε σειρά χαμηλότερο για τα τελευταία 8 ετία ποσό. Ποσοστό καλύτερα. Η πρόταση είναι οργανωμένη αντίστοιχα με αυτήν ε, τη προηγούμενη χρονιά, με βάση την πρόταση Επιτροπή των Προπολογισμών. Δηλαδή, έχουμε ε, τι τακτικέ δαπάνε και τι έκτακτε δαπάνε, οι οποίε δυστυχώ στον τομέα τη ασφάλεια χρειάστηκε να ενισχυθούν και φέτο ε, κατά 2%. Ε, 0, 2% αύξηση και γιατί το Συμβούλιο αποφάσισε να μετατραπεί σε πλήρης, πλήρους καλύψεως γλώσσα η Ιρλανδική, άρα χρειαζόμαστε και τη μετάφραση και τη διερμηνία και πρέπει να προετοιμαστούμε γι' αυτό, άρα έχουμε ένα 0,2% επιπλέον και αυτή είναι η δομή ε, την οποία έχει αποφασίσει, έχουμε αποφασίσει, έχει αποφασίσει το Κοινοβούλιο στον προπολογισμό του 2016 ήδη. Ιδιαίτερα Ωστόσο, σημαντική είναι η αύξηση όσον αφορά τον τομέα της ασφάλειας δυστυχώς ε, κοιτώντας γενικά την κατάσταση, βλέπουμε ότι γίνονται κάθε εβδομάδα επιθέσεις γύρω-γύρω από την Ευρώπη. Στην Μέση Ανατολή έχουμε πόλεμο με συμμετοχή και κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό σημαίνει μια τελείως νέα κατάσταση διακινδύνευσης που δεν φαίνεται να είναι βραχυπρόθεσμη ή περιστασιακή, δεν πρόκειται να τελειώσει μια κατάσταση την οποία θα έχουμε να ζήσουμε για τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον και επιβαρυντική συνθήκη είναι το γεγονός ότι οι Βρυξέλλες είναι μια πόλη στην οποία δυστυχώς όπως μάθαμε ε, υπάρχουν πολλοί Ισλαμιστές, άλλωστε μας το έδειξαν οι επιθέσεις στο Παρίσι. Το Κοινοβούλιο ευτυχώ από το 2009 αναλαμβάνει, ανέλαβε τακτικά και αλλεπάλληλα βήματα για τη βελτίωση της οργάνωσης της ασφαλείας Το 2009 είχαμε μια μικρή μονάδα ασφαλείας στο Κοινοβούλιο, η οποία μετετράπησε σε διεύθυνση, τώρα είναι γενική διεύθυνση. Έτσι βήμα το βήμα εγκαταλείψαμε την προσέγγιση της ανάθεσης εξωτερικές υπηρεσίες ασφαλείας, εσωτερικεύτηκε δηλαδή αυτή η υπηρεσία, έγινε ιστορική του Κοινοβουλίου, αλλά το καθοριστικό ήταν ότι ο στρατηγικό έλεγχο τη ασφάλεια μα και ο σχεδιασμό ο στρατηγικό τη ασφαλείας μα είναι πλέον στα χέρια μα, δεν, είναι, δεν ανήκει σε εξωτερικέ υπηρεσίε, αλλά σε υπαλλήλου μακροπρόθεσμα απασχολούμενο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι επιθέσει από τον προηγούμενο ήδη Ιανουάριο στο Παρίσι με το Σαρλί Εμπτό οδήγησαν σε ενίσχυση των συνθήκων ασφαλεία για τι εισόδου του Κοινοβουλίου, μια αναδιοργάνωση των συνθήκων ε, εισόδου στο Κοινοβούλιο, έτσι ώστε σε περίπτωση αντίστοιχων επιθέσεων με αυτές του Παρισιού να μην μπορούν οι τρομοκράτες να μπουν ανεμπόδιστοι ε, στα κτίρια. Οι είσοδοι λοιπόν έκλεισαν ήδη στη μεριά της πλατείας του Λουξεμβούργου και από την οδό Βίρτς ολοκληρώνται εργασίες για να παραδοθεί η είσοδος τον Απρίλιο. Το Προεδρείο έχει εξασφαλίσει την εισαγωγή για το 2017 μιας νέας ε, ασφαλούς και μη δυνατόν να πλαστογραφηθεί ταυτότητας για όσους εργάζονται εδώ και βέβαια παρακολουθούμε συστηματικά η αδίποτε ε, εναπομείναντα ε, σημεία αδύνατα στην αλυσίδα της ασφάλειας και κοιτάμε όχι μόνο τις μεγάλες εισόδους ε, και απαιτούμε βέβαια αυτές να έχουν ε, το υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας αλλά κάθε είσοδο στο κοινοβούλιο γιατί βέβαια η όποια είσοδος έχει τη λιγότερη ασφάλεια προσδιορίζει το γενικό επίπεδο ασφάλειας για όλο το κτίριο. Αυτή η δουλειά γίνεται βήμα το βήμα, το κύριο κτίριο ασφαλώς αλλά και τα περαιτέρω κτίρια, τα κτίρια του Στρασβούργου και ασφαλώς και τα νέα κτίρια όπως το ΚΑΤΖ του Λουξεμβούργου και το κτίριο Μάρτενς εκεί. Δεύτερον, υπάρχουν ε, ε, επιφάνειες με τζάμι οι οποίες δεν είναι ασφαλείς κυρίως στον, ε, στην πρόσωψη από την πλευρά του εστιατορίου, εστιατορίου και καντινα Surf self-service, αλλά και σε άλλα σημεία, μεγάλες επιφάνειες με γυαλί, οι οποίες είναι ευάλωτες σε περίπτωση επιθέσεως, γιατί το γυαλί αυτό δεν είναι ασφαλές και μπορεί να εκραγεί προς τα έσω του κτηρίου. Άρα πρέπει να ασφαλιστούν αυτές οι επιφάνειες. Ε, δυνατότητες τεχνικές υπάρχουν, τις απαληθεύουμε αυτή τη στιγμή. Επίσης θέλουμε να εξασφαλίσουμε την προστασία των κυρίων κτηρίων έναντι ενδεχόμενης επιθέσεως με οχήματα. Πέραν αυτού έχουμε να εξετάσουμε, ο αντιπρόεδρο άλλωστε Βίλαντ το ανέφερε νωρίτερα, ε, πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν και τις κύριες ε, προσβάσεις στο χώρο στα κτίρια τη ολομέλεια, οδού Βίρτ και Βοτ και εάν αυτές μπορούμε να τις αποκλείσουμε από την οδική κυκλοφορία ή αν μπορούν να μετατραπούν σε πεζοδρόμους, Φερρυπίν. Εδώ έχουμε να κάνουμε με συζητήσεις εν εξελίξη με τις αρχές του Βελγίου. Προβλέπεται το Μάρτιο συνάντηση. Οι αντιπρόεδροι Βίλαντ και Σασόλη θα αναλάβουν αυτές τις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με τις βελικές αρχές. Από τον Ιανουάριο επίσης έχουμε εξωτερική προστασία από τις βελγικές αρχές που προσφέρει, προσφέρουν ένοπλη προστασία. Ενισχύεται δε αυτή και κοιτάμε να εξασφαλίσουμε και χώρους διαμονής, ε, φυλάκια για τους φρουρούς αυτούς. Η υπηρεσία οδηγών τώρα ήταν ένα άλλο θέμα, το οποίο με έχει απασχολήσει, το έχω συζητήσει εντατικά με τον ε, πρόεδρο, με τον αντιπρόεδρο, έχει συζητηθεί και στο Προεδρείο. Δεν έχουμε καταλήξει σε καμία απόφαση. Ο Πρόεδρος παρακάλεσε μόνο το θέμα να μπει στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδριάσεως του Προεδρείου για τις 7 Μαρτίου συγκεκριμένα. Ωστόσο θεωρούμε πως για λόγους ασφαλείας αλλά και για να έχουμε μια ε, ορθολογική επάνδρωση της υπηρεσίας. Είναι σκοπιμότερη η εσωτερική οργάνωση της υπηρεσίας των οδηγών. Ένα δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο είναι οι γλώσσες. Τα ιρανδικά τώρα μετατρέπονται σε γλώσσα σε πλήρη ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, και ίσως να μην είναι γνωστό τη Σπάσιν ακόμη, Επιπλέον ε, όμως ε, βρίσκονται εν εξελίξει οι οι συζητήσεις μεταξύ της ε, Κυπριακής Δημοκρατίας της Κύπρου και του τουρκικού τμήματος στο νησί. Είναι κάτι το οποίο είναι να εξελίξει, δεν μπορούμε βέβαια να προεξοφλήσουμε επιτυχία έκβαση σύντομα, αλλά υπάρχει μία ελπίδα πως μπορεί να υπάρξει συνεννόηση σύντομα και έτσι να γίνει η επανένωση της Κύπρου σε ορατό μέλλον. Αυτό βέβαια θα σήμαινε πως και η γλώσσα της Βόρειας Κύπρου, τα τουρκικά δηλαδή, θα μπορούσαν να προσφερθούν από τις υπηρεσίες μας, ανεξαρτήτως βεβαίως και των συζητήσεων για την ε, λύση του Κυπριακού και την επανένωση του νησιού. Θα είχαμε δηλαδή 25 γλώσσες στο Ευρω... Ε, ανάλογα και με τις εξελίξεις και την επανένωση στην Κύπρο, θα είχαμε 25 λοιπόν ε, γλώσσες. Ε, βλέπω εδώ την έκθεση του εισηγητού για την αναδιοργάνωση των γλωσσικών μας υπηρεσιών. Έχουμε καταβάλει από τον τελευταίο χρόνο πολύ μεγάλες προσπάθειες για την αναδιοργάνωση όχι μόνο της ερμηνείας αλλά και της ε, μετάφρασης. Κοιτούμε να οργανωθούμε με βάση τη ζήτηση, αλλά θα χρειαστεί περαιτέρω μεταρρύθμιση για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε όπως το θέλουμε, μακροπρόθεσμα, την πολυγλωσία. Και αυτό θα χρειαστεί προσπάθειες από όλους. Για τα κτίρια έχουμε μία σειρά σχεδίων για κτίρια. Ένα νέο κτίριο του CAD, Κόνραντ Αντενάουερ του Λουξεμβούργου, που προχωρεί ταχαίως. Το Προεδρείο το προηγούμενο καλοκαίρι με δική μου πρόταση αποφάσισε ο, ε, να μην περιοριστεί ο όγκος του κτηρίου έτσι μειώνεται το κόστος κατά 50 εκατομμύρια, η εκτίμηση του κόστους κατά 50 εκατομμύρια ευρώ και έτσι μπορούμε στο Λουξεμβούργο να έχουμε την ίδια κλίδα τετραγωνικών μέτρων, 11 δηλαδή τετραγωνικά ανά ε, εργαζόμενο στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο. 11 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό σημαίνει, με τη βάση αυτή, ότι μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες των 2.400 εργαζομένων μονίμων υπαλλήλων και 600 εξωτερικών συνεργατών του Λουξεμβούργου, να τους εξασφαλίσουμε τους χώρους εργασίας και με περιορισμένη ε, δαπάνη, περιορισμένη κατά 50 εκατομμύρια ευρώ, περιορίζοντας αυτόν τον όγκο του κτηρίου. Εάν περαιτέρω χρειαστεί να επεκταθεί το κτίριο, αν υπάρξει ανάγκη δηλαδή για νέα εγκαταστάσει ή για περισσότερε εγκαταστάσει, είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποφασίσει η προσεχή σύνθεση του Κοινοβουλίου μετά τι εκλογέ. Θα ήταν λάθο πάντω τώρα να λαμβανόταν απόφαση για εγκαταστάσει κτηριακέ οι οποίε δεν χρειάζονται. Το κτίριο Μάρτεν στι ε, Βρυξέλλε ακολουθεί το χρονοδιάγραμμα που έχει οριστεί. 1η Απριλίου του 2016 θα παραδοθεί ε, στο σύνολό του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ακολουθήσουν δύο έτη για την εσωτερική προσαρμογή των χώρων, να ανοίγει στις 16 ε, Νοεμβρίου. Το πλαίσιο των δαπανών έχει τηρηθεί όπως είχαμε συμφωνήσει και με την Επιτροπή των Προϋπολογισμών. Θα υπάρξουν σε κάποια σημεία ε, αυξημένες δαπάνες στο χώρο της ασφάλειας συγκεκριμένα, γιατί με τις νέες συνθήκες και προϋποθέσεις ε, αποφασίστηκε ότι θα χρειαστεί να εγκατασταθεί η υπηρεσία ελέγχου στις εισόδους, ελέγχου ασφαλείας στις εισόδους, κάτι που δεν είχε αρχικά προβλεφθεί. Η Επιτροπή συμμετέχει με 800.000 ετησίως στη χρηματοδότηση για τον οίκο της Ευρωπαϊκής ιστορίας. Ε, καλύπτει λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Δαπάνες που αφορούν και τους επισκέπτες για το Άτριουμ. Από το Σεπτέμβριο φέτος θα είναι διαθέσιμη η πρόσβαση και σε ε, λεωφορεία επισκεπτών και θα υπάρχει δυνατότητα να προσέρχονται σε συνομιλίες με βουλευτές οι ε, επισκέπτες ο σταθμός, ο στερεοδρομικός σταθμός Λουξεμβούργου κλείνει και ελπίζουμε ότι θα ξανανοίξει εγκαίρως για την παράδοση του οίκου ε, της ευρωπαϊκής ιστορίας. Επομένως όλα αυτά πλέον για το 2017 δεν θα έχουν επίδραση στον προπολογισμό. Επίσης το 2016 κλείνει το ζήτημα της ανακαίνησης του κτηρίου Χάβελ με 300 περίπου νέες ε, εγκαταστάσεις και γραφεία για τους βουλευτές και θα έχουμε τη δυνατότητα για ένα μίνι μίνι-παρλαμεντάριο στο ε, Στρασβούργο που θα ανοίξει το 2017 και ένα ακόμα μίνι μίνι-παρλαμεντάριο στο Βερολίνο που θα ανοίξει μέσα στο 2016. Δηλαδή το 2016 είναι ένα έτος μέσα στο οποίο ε, ολοκληρώνονται διαδικασίες που έχουν αποφασιστεί τα τελευταία χρόνια και έτσι μέσα στο 2017 θα δούμε μια σημαντική αλλαγή και ε, αποφόρτιση στον προϋπολογισμό. Πολύ σωστά επισημαίνει ο εισηγητής βεβαίως ότι παρόλα αυτά χρειάζεται μια μεσοπρόθεσμη στρατηγική κτίρια εκεί που ίσως έχει ε, λιγότερη ε, σημασία η επιβάρυνση για την τρέχουσα θητεία, αλλά ξέρουμε όλοι ότι τα κτηριακά ζητήματα είναι, ζητήματα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός, οι συμβάσεις, οι αναθέσεις Επομένως, εάν θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να λάβει αποφάσεις στο επόμενο κοινοβούλιο, κατά την επόμενη θητεία, θα πρέπει να έχουμε μια μέσο πρόθεσμη κτηριακή στρατηγική, η οποία θα έχει κάνει σχετική παρασκευαστική, προπαρασκευαστική δουλειά εγκαίρως. Ένα προσχέδιο λοιπόν κατατέθηκε το Σεπτέμβριο του 2015 στο Προεδρείο με κέριο ζήτημα τις ανάγκες ανακαίνησης του κτηρίου PHS του Polaris Το ανέφερε ο κύριος Βίλαντ μόλις τώρα. Και το θέμα είναι σε τι επίπεδο φιλοδοξίας θέλουμε να αρθούμε για την ανακαίνιση αυτή. Ένα στοιχείο το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να λάβουμε υπόψη είναι και να κρίνουμε εάν και τι ανάγκες έχουμε μέσω και μακροπρόθεσμα για τις γλώσσες. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο μία αίθουσα που να καλύπτει και τις 24 γλώσσες στις 24 καμπίνες. Οι άλλες αίθουσες έχουν το πολύ 19 γλώσσες δυνατότητα να καλύψουν. Άρα και έχουμε δεσμευθεί για την πολυγλωσσία, την κάλυψη όλων των γλωσσών Ούτε και πρόκειται βέβαια να υποχωρήσουμε. Ε, δεν είναι το πρόβλημά μα δηλαδή ότι δεν έχουμε αρκετά χρήματα ή ότι δεν μα φτάνουν οι διερμηνεί. Αλλά δεν έχουμε τι υποδομέ, τι τεχνικέ υποδομέ να υλοποιήσουμε αυτή τη δέσμευση που έχουμε αναλάβει. Δηλαδή να εξασφαλίζουμε για τον κάθε βουλευτή στη γλώσσα του τη γλωσσική υπηρεσία που χρειάζεται. Πέραν αυτού και επιπλέον, εάν κοιτάξουμε και το ζήτημα της Κύπρου που έθιξα, η εξελίξεις που αφορούν ε, περαιτέρω υποψήφιες χώρες, Σερβία, Βοσνία, Αλβανία, Μακεδονία, Μαυροβούνιο, ήδη υπάρχουν υποψήφια κράτη τα οποία θα μας οδηγούσαν με την ένταξή τους στις 30 γλώσσες. Αν λοιπόν θέλουμε να συνεχίσουμε το υφιστάμενο καθεστώ πολυγνωσία, τη δυνατότητα δηλαδή για τον κάθε βουλευτή να εργάζεται πράγματι στη γλώσσα του και, όχι, και να μην βρίσκεται αυτό το δικαίωμα μόνο επί χάρτου, τότε θα πρέπει να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα πώς εξασφαλίζουμε την, τις υποδομές σε χώρους, σε αίθουσες, έτσι ώστε να μην παραμένει το δικαίωμα αυτό επί χάρτου, αλλά πράγματι να ε, υλοποιείται. Σας ευχαριστώ. Merci, Ευχαριστούμε, κύριε Γενική Γραμματέα. Τώρα, θα ακούσουμε τους σκιώδεις εισηγητές, αν θέλουν να πάρουν το λόγο. Ο κύριος Ρίμπιχ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ επακριβής η τοποθετήση σας και πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται ενώπιον νέων προκλήσεων, ιδιαίτερα στο θέμα της ασφάλειας. Την τελευταία ανάλυση αποφάσει που παίρνουμε έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των συναδέλφων μας για τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες, μήνες και χρόνια ακόμη. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα να αναπτύξουμε τη δική μας στρατηγική, να δούμε τι χρειαζόμαστε και σε επίπεδο προσωπικού, να έχουμε στο δυνατόν ε, αυτοματοποιημένους ελέγχους ασφαλείας με το face detection αναγνώριση, δηλαδή χαρακτηριστικών προσώπου, για το ποιος μπορεί να μπαίνει χωρίς περαιτέρω έλεγχο στο κοινοβούλιο. Στην Αυστραλία, παραδείγματι, στο αντίστοιχο κοινοβούλιο έχουν ε, οι υπάλληλοι ασφαλείας στο κουβούκλιο που κάθονται μια οθόνη στην οποία βλέπουν αμέσως την απεικόνηση του προσώπου όποιου εισερχομένου στο κτίριο. Είναι κάτι το οποίο πιστεύω θα μπορούσε να μας απασχολήσει γιατί θα εξασφάλιζε μια πρόσκοπτη ε, δυνατότητα εισόδου για το προσωπικό του συνεργάτε μας και όσους δουλεύουν τακτικά στο κοινοβούλιο δηλαδή, από τις εισόδους. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να σα απασχολήσει όχι μόνο για τι Βρυξέλλε και το Στρασβούργο, αλλά και για το Λουξεμβούργο. Πρέπει να γίνει σχετική προσαρμογή των κτηρίων. Και αυτό θα πρέπει να μα απασχολήσει με την έννοια του τι είδου ε, ε, λογική πρέπει να ακολουθήσουμε στην υπόθεση αυτή, ώστε να έχουμε ισοδύναμα μέτρα ασφαλεία και, και στι τρει έδρε και για τι ε, γλωσσικέ τεχνολογίε ασφαλώ. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια δυνατότητα να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητά μας αν τις αξιοποιούσαμε με αυτοματοποιημένες υπηρεσίες για διάφορες ε, συναντήσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ποιότητα των συναντήσεων. Επίσης έχουμε αποφασίσει όλοι τα δημόσια κτίρια να βελτιώσουν την ενεργειακή τους αποτελεσματικότητα κατά 3%. Είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη στα σχέδιά μας. Το έχουμε αποφασίσει εμείς και πρέπει να το υλοποιήσουμε και στα δικά μας κτίρια. Και αναλόγως εξοικονομούμε και πόρους με την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ενεργειακής των κτιρίων μας. Μακροπρόθεσμα. Μπορούμε λοιπόν να το ε, εξασφαλίσουμε αυτό. Για το του Ταράντ. Θέλω να πω ότι η επιθυμία του για την εγκατάσταση της ε, Ένωσης Παλαιών Βουλευτών στο Στρασβούργο όπου θα μπορούν να συνευρίσκονται οι παλιοί βουλευτές ε, χωρίς περιορισμούς, χωρίς όρια είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να εξασφαλιστεί εάν ε, βρίσκαμε λύσεις για την λειτουργία των κτηρίων ε, με εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται ήδη, τους επισκέπτες ε, και ιδιαίτερα από την περιοχή γύρω από την Αλσατία που επισκέπτονται τα κτίρια τακτικά. Είναι κάτι το οποίο λοιπόν μπορούμε να προβλέψουμε σε όρους τακτικούς, γιατί δεν θέλουμε να αποτελούμε ξένο σώμα στο ε, Στρασβούργο, αλλά να είμαστε παρόντες διαρκώς στις δραστηριότητες. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα λάβουμε θετική ανταπόκριση από τις πολιτικές ομάδες στην πρόταση που έχουμε αποστείλει. Η Ένωση αυτή των παλαιών βουλευτών έχει και μια πολύ σημαντική κοινωνική διάσταση σε σχέση με την ε, κρίση που αντιμετωπίζουμε την εποχή αυτή είναι πολύ σημαντικά τα εξή δύο. Η επικοινωνιακή πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εάν δούμε τι είδου αποπληροφόρηση ε, διαδίδεται από διάφορες ε, οντότητες και μονάδες εκτός και εντός Ευρώπης, μη κυβερνητικές οργανώσεις κτλ. Παραπληροφόρηση λοιπόν και νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον των πολιτών Όλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βελτιώσουμε την ε, επικοινωνιακή μας πολιτική και την ενημέρωση για τις δραστηριότητε μας. Ιδιαίτερα λοιπόν θα μπορούσαμε να προβλέψουμε ένα σύστημα κατάρτισης νεαρών δημοσιογράφων, ενημέρωσης τους ώστε να γνωρίζουν, να εξοικειωθούν περισσότερο με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να μπορούν να τις παρακολουθούν και να αντιλαμβάνονται την, ε, το πλέγμα αυτό της κοινοβουλευτικής δουλειάς κατά τρόπο πιο διαφανή. Και νομίζω ότι ένα κέντρο μέσων μαζικής ενημέρωσης και κατάρτισης δημοσιογραφικής θα μπορούσε να αποτελέσει ακριβώς σε περίοδο κρίσης ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο ώστε να βελτιωθούν οι δυνατότητες επικοινωνίας με τους πολίτες και μέσα βεβαίω και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των βουλευτών. Αυτά είναι τα σημαντικότερα σημεία από δική μας πλευρά Ευχαριστούμε κύριε Ρουμπίκ. Ο κύριος Σοντελανό τώρα από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίαση και του Αντιπροέδρου και του Γενικού Γραμματέα. Οι πληροφορίες αυτές που μας έδωσαν είναι σίγουρα πολύ ενδιαφέρουσες. Ευχαριστώ και τον εισηγητή, ο οποίος παρουσίασε τις προτάσεις του όσον αφορά την ασφάλεια, τα νέα κτίρια, νέες γλώσσες, υπηρεσία οδηγών κλπ. κλπ. Αυτό που θέλω όμως να προσθέσω είναι ότι αυτός ο προπολογισμό, ακόμα και αν περιορίζεται κάτω από 20% από το συνολικό προϋπολογισμό, βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Ευρωπαίων πολιτών και των δημοσιογράφων. Το ξέρουμε εμείς αυτό. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικοί και πάρα πολύ συγκεκριμένοι στο τι θέλουμε να κάνουμε. Αυτό λοιπόν που προσέχουμε εμείς οι σοσιαλιστές είναι αύξηση 3,9% ενώ ο πληθωρισμός ανακοινώνεται στο 1,7% αλλά εγώ δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι το επίσημο νούμερο γιατί υπάρχουν χώρες όπου ο πληθωρισμός είναι 0% και διαμαρτυρόμαστε. Λέμε ότι δεν τα καταφέρνουμε να ανεβάσουμε τον πληθωρισμό στο επίπεδο του 2% που θα ήταν το ιδεώδες. Οπότε πρέπει να αναρωτηθούμε για αυτά τα στοιχεία. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα. Ποιο είναι ο πραγματικό πληθωρισμό τη Ευρώπη σήμερα. Θα ήθελα να ξέρω περισσότερα από αυτού. Έπειτα διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν γραμμές με μεγάλη αύξηση. Τι κτίζουμε, για παράδειγμα, η ασφάλεια. 31% αύξηση στην ασφάλεια. Έτσι έρχομαι στο θέμα της ίδιας της δομής του προπολογισμού που δεν περιλαμβάνει τμήμα επενδύσεις εγώ δεν είμαι συνηθισμένο σε κάτι τέτοιο. Στις δικές μου τοπικές αρχές λειτουργούμε αλλιώς. Μπορούμε δηλαδή με τα έξοδα λειτουργίας να χρηματοδοτήσουμε και επενδύσεις. Ίσως θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό περισσότερο. Θα ήταν χρήσιμο εξάλλου προκειμένου να προβάλλουμε προς τα έξω τους λογαριασμούς του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Για το θέμα της ασφάλειας των κτηρίων δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Όλοι τη θέλουμε αλλά να καταλάβουμε καλύτερα πώς λειτουργούν τα πράγματα, τι μελέτες έχουν γίνει, ποιοι εμπειρογνώμονες ε, γνωμοδότησαν, τι προτάσεις υποβλήθηκαν. Θα θέλαμε δηλαδή να ξέρουμε ποιο είναι το σχέδιο όσον αφορά την ασφάλεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί τότε θα καταλάβουμε καλύτερα τι πρέπει να κάνουμε και τα επόμενα χρόνια. Αναφερθήκατε στη, στα τζάμια, τις μεγάλες επιφάνειες με τζάμια που αποτελούν δυνάμει κίνδυνο, τζαμαρίες. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω περισσότερο τι τεχνικές έχετε αποφασίσει να χρησιμοποιήσετε. Είναι αλήθεια ότι 15 επιπλέον εκατομμύρια ευρώ χρησιμοποίησαμε πέρυσι. Έτσι θα συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια. Ας προσπαθήσουμε να διακανονίσουμε λίγο αυτό το ζήτημα. Τώρα, όσον αφορά τους οδηγούς, την υπηρεσία οδηγών και κατά πόσο θα επανδρώνεται εκ των έσω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εδώ χρειαζόμαστε περισσότερες διευκρινήσεις. Τι κρύβεται θα μπορούσα να πω ή τι μπορεί να προσφέρει επιπλέον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους Ευρωβουλευτές και τι θα γίνει με τους οδηγούς, γιατί πρέπει να έχουμε υπόψη μας τι θα τους προτείνουμε, θα είναι οδηγοί, θα έχουν και άλλα καθήκοντα, ε, θα... τι γίνεται με την κατάρτιση. Είναι και αυτά ερωτήματα να αποφασίσουμε για μια αλλαγή στην υπηρεσία αυτή. Όσον αφορά τώρα την βοήθεια εξαγουλευτών. Με τη μείωση της χρήσης του χαρτιού είναι αλήθεια ότι η πληροφορική μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και να περιορίσει τη χρήση του χαρτιού. Ναι, όμως, θα έπρεπε να δούμε τι χρήματα πηγαίνουν και εκεί υπάρχουν κονδύλια στους βουλευτές για τέτοιους σκοπούς. Αυτό που θα ήταν ενδιαφέρον είναι να δούμε την πρόσβαση στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από την εκλογική μας περιφέρεια. Αυτό θα ήταν ενδιαφέρον. Για τις υπηρεσίες έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αναγκαίο να προωθήσουμε περισσότερο την ποιότητα και όχι την ποσότητα. Σίγουρα ακαδημαϊκές έρευνες βοηθούν τους ευρωβουλευτές στο έργο τους. Αλλά όσο περισσότερους συνομιλητές έχουμε τελικά καταλήγουμε σε ένα μπέρδεμα και δημιουργείται σύγχυση για τους ίδιους τους ευρωβουλευτές. Και εδώ λοιπόν θα θέλαμε κάποια διευκρίνηση για τον ρόλο που έχει ο καθένας στο τομέα της έρευνας. Και έρχομαι τώρα στην επικοινωνία και την ε, συγκέντρωση των ε, γραφείων Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις ε, πρωτεύουσε. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά καλό θα ήταν να γίνει. Είμαστε Πάντως για το μίνι παρλαμεντάριουμ Βρυξέλλες είπατε θα έχει και στο Στρασβούργο και στις 9 Μαΐου είπατε θα γενιάσουμε και αυτό στο Βερολίνο. Μήπως θα πρέπει να σταματήσουμε τις δαπάνες ή να ζητήσουμε από τις χώρες μέλη αν θέλουν να αναλάβουν εκείνες τη δαπάνη. Τώρα για τις ε, διάφορες προτάσεις που γίνονται, τα διάφορα για τις καντίν τις λεγόμενες, τα μεταλλικά δηλαδή κυβότια τα οποία για να έρχονται Βρυξέλλες, Στρασβούργο, Στρασβούργο, Βρυξέλλες. Μου λένε ότι είναι τεράστια δουλειά, ότι είναι ένα σωρό φορτηγά τα οποία πηγαίνουν και έρχονται. Ε, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν είναι δυνατόν να μειώσουμε τα πράγματα που μεταφέρονται έτσι. Θα μπορούσαν και εδώ να γίνουν οικονομίες, να μοιράζονται πολύ πάλι το ίδιο μεταλλικό κυβότιο. Όπως και το θέμα των αυτοκινήτων, των οχημάτων. Φυσικά και είμαστε υπέρ να κοιτάξουμε το θέμα των ηλεκτρικών οχημάτων, ιδιαίτερα για μικρές ε, αποστάσεις από το σταθμό στο κοινοβούλιο, στο κτίριο. Θα ήταν πολύ έξυπνο να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτρικά οχήματα για τέτοιες μικρές αποστάσεις. Με απασχολεί και το θέμα των ταξιδιών των Ευρωβουλευτών. πώς θα μειωθεί το κόστος. Να το σκεφτούμε, ναι. Όπως το προτείνετε, αλλά εξαρτάται ποια. Τα μικρά ταξίδια. Δεν υπάρχει εκεί ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά αν πρέπει να πάμε σε μεγαλύτερες, σε πιο μακρινές αποστάσεις, να το κοιτάξουμε, αλλά να έχουμε και υπόψη μας ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον παράγοντα άνεση. Αυτές, Πρόεδρε, είναι οι παρατηρήσει μου και άλλοι θα έχουν παρατηρήσει σίγουρα, συνάδελφοι. Τέλος, θέλω να στηρίξω την ιδέα ότι πρέπει να διατηρήσουμε την πολυγλωσία, ακόμα και αν κοστίζει. Είναι κομμάτι του ίδιου του DNA της Ευρωπαϊκής Ένωσης η πολυγλωσία. Αν τα τουρκικά προσθεθούν, εντάξει, στο κάτω-κάτω θα είναι καλό νέο για την Κύπρο αυτό. Οπότε, ναι, δεν πρέπει να τσιγκουνευόμαστε εδώ όσον αφορά την πολυγλωσία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε από το ECR τώρα. Α, δεν είναι εδώ γιατί ο συνάδελφο μάλλον είναι στον Εμένο Βασίλειο λόγω τη επικαιρότητα. Ο κύριο Στόρβαλτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να σας πω το εξή. Να σας μιλήσω στα αγγλικά, γιατί θα, σας μιλήσω κάποια γλώσσα που δεν είναι ούτε φιλανδικά, ούτε σουηδικά η μητρική μου γλώσσα, αλλά ούτε και τα Ιρλανδικά. Ε, σύντομα σχόλια και όσα ακούσαμε για την ε, μετάφραση είχα να σας πω. Έχω κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά τα ποσά για το ε και για το h. 4,3 100% και επίσης θα πρέπει να είναι 62 τα εκατομμύρια αλλά περιμένω να μου το διευκρινίσετε. Επίσης θα πρέπει να διαχωριστεί το θέμα της ε, αύξησης των δαπανών της ε, ασφάλειας από το θέμα της Ιρλανδικής γλώσσας. Επίσης μου φάνηκε ελαφρώς άστοχο το να ζητηθεί από τον ε, κύριο Γενικό να έρθει σε επαφή με τους Ιρλανδούς συναδέλφους για να υπάρξει κάποια εκλογήκευση. Αυτό. Η αντιστοιχή σε εκείνο που είχε πει πριν από τρει αιώνε ο Γκρέμ Σουίφτ, τότε που είχε υπάρξει ο μεγάλο λοιμό στην ε, Ιρλανδία και είπε ότι μια που δεν έχουν τι να φάνε, α φάνε τα παιδάκια του, τα μωρά του. Οπότε Α δούμε υπ' αυτό το φως, με, αυτό το πνεύμα. Έχουν περάσει πολλά χρόνια, λέει ο Και νομίζω ότι έχω ξανασκεφτεί το τι γίνεται όσον αφορά τις εκλογικές μας ε, περιφέρειες. Νομίζω πρόκειται για κάποιες νέες διατάξεις, ε, κάποιοι ερχόμαστε από συνεδριάσεις, εγώ έρχομαι από μια περιοχή όπου θα πρέπει από το Ελσίνκι μέχρι το Όκι να κάνουμε απόσταση 1300 ε, χιλιόμετρων. Στο Λουξεμβούργο κάποιος που πηγαίνει μάξιμο 80 τόσα χιλιόμετρα μα θέλει να πάει στο πιο μακρινό σημείο που είναι η εκλογή του περιφέρεια ας πούμε. Οπότε θα πρέπει αντιστοίχως να γίνει και η προσαρμογή και η ρύθμιση σχετικά με αυτό. Οπότε και ο απολογισμός σε σχέση με τα οδηπορικά μας δεν είναι θέμα ψηφιοποίηση για την οποία γίνεται πολλή κουβέντα. Αλλά θα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση που ίσως να μην αφίσταται τόσο πολύ του, χαρτιού της εφεύρεσης του Κοντεμβερή. Τέλος πάντων, Τώρα όσον αφορά τα κτίρια. Σύμφωνα για το παρλαμεντάριο και το μίνι παρλαμεντάριο όπως προαναφέρθηκε. Αν θέλετε να φτιάξετε μίνι παρλαμεντάρια σε όλα τα κράτη-μέλη, ε, τότε θα πρέπει αυτός που θα τον λάβει να κλείσει μια θέση στο τρελοκομείο. Τώρα όσον αφορά τους ε, οδηγούς του σοφέρ δεν είμαι και τόσο ενθουσιασμένος με την ιδέα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Από ό,τι γνωρίζω, τα Τέσλα είναι αρκετά ακριβά. Άρα δεν είναι αυτή η λύση στο πρόβλημά μας. Αυτό είναι μάλλον για να δημιουργήσει εντυπώσει ότι δηλαδή ότι είμαστε ε, περιβαλλοντικών λύσεων. Μιλήσατε και για τα μπαούλα αυτά τα κουτιά που μεταγίνονται πάνω στο Στρασβούργο. Ας δούμε όμως την ουσία του θέματος. Ας δούμε δηλαδή, όχι το θέμα των μπαούλων για το Στρασβούργο, για το ίδιο το Στρασβούργο γιατί πρόκειται για, για απίστευτη δαπάνη, απίστευτη διασπάθηση. Κατά τα άλλα πάντως νομίζω ότι ο συνάδελφος με την έκθεσή του επετέλεσε πάρα πολύ σωστό έργο και νομίζω ότι όταν ε, μπουν οι τελευταίες πινελίες θα είναι υπέροχη έκθεση. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε και τώρα. Το λόγο έχει ο κύριος ο Μαρζή, ο οποίος φαντάζομαι θα μας πει πόσο ενθουσιασμένος είναι για την πρόταση που αφορά τα Ιρλανδικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Γενικέ, λέει ο κύριος Ομαρζή, όσον αφορά το σχέδιο προβλήματο του Κοινοβουλίου, είναι κάποιο λεπτό θέμα το οποίο θίγουμε. Αυτό είπατε κι εσείς για την ασφάλεια του προσωπικού ε, και για το, το, το Είναι θέμα του καταστατικού που διέπει το προσωπικό. Επίσης είναι και θέμα συνθήκων εργασίας των βουλευτών. Και σας τονίζω ότι δεν μπορώ να λησμονήσω ότι αυτή μας η συνεδρίαση μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Παρά την πρώιμη φάση των συζητήσεων. Έγινε μια πρώτη συζήτηση με τους ε, σκιώδεις εισηγητές που συναντήσαμε τον ε, εισηγητή μας. Ήταν πάρα πολύ μεστή αυτή η συνεδρίαση, αυτή η συζήτηση και εκεί πέρα ανεβήθησαν πολλά ερωτηματικά. Οφείλω να σας πω ότι δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα πρέπει εδώ και τώρα, σήμερα, να βγάλουμε τα άπλυτα στη φόβρα όσον αφορά τα, ερωτηματικά, ας πούμε, για την ασφάλεια. Και Επίσης για το κατά πόσον σεβόμαστε το προσωπικό, αν συζητήσουμε έτσι ανοιχτά την δημιουργία της συνεργασίας, κατάργηση της συνεργασίας, αν συζητάμε επίσης για το καταστατικό που διέπει το προσωπικό. Ούτε νομίζω ότι εδώ είναι το κατάλληλο βήμα για να μπούμε στις λεπτομέρειες όσον αφορά τις ε, συνθήκες εργασίας των ε, Ευρωβουλευτών για τα, τα διάφορα κονδύλια, τις τυχόν αυξήσεις κλπ. Οπότε και αυτό και εγώ επιφυλάσσομαι και θα σας πω τις παρατηρήσεις μου στην επόμενη συνάντηση ό,τι κανονιστεί μεταξύ ημών και του Προεδρείου του Κοινοβουλίου. Οπότε τώρα δεν θέλω να αναλωθώ σε πράγματα πολιτικά Ο κύριος Βαλή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το κείμενό του. Πολλά είναι τα ενδιαφέροντα σημεία τα οποία μπορούν να είναι βάση συζητήσεων και θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε πίεση από τα ΜΜΕ παντού στα θεσμικά όργανα και ιδίως στο Κοινοβούλιο έχουμε το ζήτημα του Brexit το οποίο το κουβεντιάζουν όλοι Οπότε η αύξηση των δαπανών για το κοινοβούλιο σημαίνει ότι ρίχνουν νερό στο μήλο αυτών που θέλουν να στείλουν τέτοια μηνύματα για δαπάνες. Οπότε βλέπουμε ότι αναφερούν τις δαπάνες τους άλλοι πολύ, άλλοι λίγο στα κρατή μέλη. Οπότε σίγουρα είναι μια δύσκολη συγκυρία και όλοι μας θα πρέπει να συγκρατήσουμε τις δαπάνες. Επίσης ε, έχουμε το 1,7% για τον πληθωρισμό. Εγώ νομίζω ότι ε, αυτό είναι δημιουργική στατιστική από της Κομισιόν και μάλλον από πληθωρισμό έχουμε σε διάφορες ε, χώρες. Άρα επομένως δεν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτά τα στοιχεία. Επίση δεν θα πρέπει να κρυβόμαστε ε, πίσω από το 20% του πέμπτου τομέα, του πέμπτου κεφαλαίου, γιατί όπως έγινε και πέρσι και φέτος θα έχουμε μια σημαντική αύξηση. Πάμε για το 2% για την ασφάλεια και επίσης το 0,2% για τα Ιρλανδικά και είπαμε ότι όλα αυτά ε, ε, δράζονται στο 1,7 το δίθεν ακόμα του πληθωρισμού και οπότε και έτσι πάμε στο 3,9 και τα 70 εκατομμύρια. Άρα δεν θα πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο παρά μόνο να κάνουμε κάποια εκλογήκευση των ε, δαπανών. Και θυμάμαι ότι πέρσι σε παρόμοια συζήτηση θέλαμε να εκλογικεύσουμε κατά 10-11 εκατομμύρια τις δαπάνες οπότε μακάρι να μπορέσει η γραμματεία με κάποια μεθοδική δουλειά να μπορέσει να εξοικονομήσει κάποιους ε, πόρους. Όσον αφορά τώρα τις ε, δαπάνες για το προσωπικό, συμφωνώ με την παραγραφό 21 της έκθεσης όσον αφορά τις γενικές δαπάνες και ίσως θα, θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την αποζημίωση για τα οδηπορικά, για αυτά τα, χιλιόμετρα που αναφέρονται. Θα πρέπει να γίνει εκ νέου υπολογισμός. Ε, επίσης θα πρέπει να αναζητηθούν οι πόροι για τις αναγκαίες δαπάνες, ούτως ώστε να δείξουν στον κόσμο ότι έχουμε θέληση να περικόψουμε τα έξοδα και των ευρωβουλευτών. Και βέβαια έχουμε το θέμα των επιδομάτων, των, των γενικών λεγόμενων επιδομάτων, που συζητήθηκαν και πέρσι. Ε, επίσης έχουμε αυτές τις υπηρεσίες ε, της μεταφοράς από τα αεροδρόμια κλπ. Ε, δεν ξέρω μήπως θα πρέπει να πληρώνουμε ένα παίρνουμε ένα ταξί. Οπότε θα μπορούσε να καλύψει το κοινοβούλιο αυτή την ανάγκη προς τα μέλη. Επίσης και για τους δρόμους μου λένε ότι με το, με το, τρένο μπορεί να μου κάνει 10-15 να πάει στο αεροδρόμιο ενώ γίνει που είστε στις Βρυξέλλες θα αργήσει περισσότερο το αυτοκίνητο τώρα όσον αφορά τα εισιτήρια για τις ε, ε, αποστολές και για το πήγαινε έλα στην χώρα μας και εδώ θα πρέπει να αποφύγουμε τα πολλά ταξίδια στην ε, business, στη διακεκριμένη θέση Και οπότε και εδώ θα δώσουμε το παράδειγμα προς και να μην δίνει τέτοια εισιτήρια ε, το γραφείο ταξιδίων. Και άρα σαν πρώτη επιλογή να δίνει εισιτήρια στην τουριστική θέση το, ε, το γραφείο ταξιδίων. Μιλάμε για πολλά εκατομμύρια που θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε για όλα αυτά τα ε, έξοδα που δεν δικαιολογούνται. Αυτό αφορά και τα μπαούλα που κουβαλάνε τα πράγματα στο ε, Στρασβούργο. Υπάρχει και την πρωτοβουλία του Αντιπρόεδρου Σασόλη. Και προσωπικά είπα ότι δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτά τα ε, μπαούλα και κουβαλάω τα έγγραφά μου. Ακριβώς αυτό το έκανα για να αποδείξω το ότι θέλουμε να ε, υπάρχει η χρήση αυτών, να περικοπεί η χρήση αυτών των ε, ε, μπάουλων όσον αφορά την ενιαία, τη μοναδική έδρα. Είδατε τι έγινε με τις δαπάνες σε σχέση με το Brexit. Τώρα όσον αφορά τα 60 εκατομμύρια για τα κόμματα ετησίως και αυτό είναι υψηλό ποσό θα μπορούσαμε και εδώ να κάνουμε περικοπές, μπορούσαμε και εμείς να ε, κάνουμε κάτι σαν βουλευτές, αλλά και η Ένωση των πρώην βουλευτών. Και άλλα θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Επίσης κάτι για τον κύριο Γενικό. Τι είναι το παραμετάριο μου στο Βερολίνο. Ε, ποιες βάσεις ξεκινήσατε την πρωτοβουλία να γίνει αυτό και, και ποιο θα είναι το κόστος, ποια θα είναι η προσθέμενη αξία του να γίνει κάτι τέτοιο στο Βερολίνο. Γιατί στο, στο Βερολίνο, καταλαβαίνω, για εξέλιξη στα σβούλα, γιατί εκεί. Καλώς, τελευταίος. Ο κύριος Ζολτέκ από τους κοιόδης εισηγητές. Α, δεν είναι εδώ όμως. Ωραία, να διευκρινίσω ότι ο εισηγητής μας ο οποίος σέβεται το χρόνο και το χρόνο ομιλίας, είχε θεωρήσει ότι ε, σε, μια μισή ώρα θα είχαμε ολοκληρώσει τη συζήτηση. Ο συγητής λοιπόν, ο κύριος Ταραντ, πρέπει να φύγει οπωσδήποτε στις 4.30 γιατί πρέπει να πάρει αεροπλάνο. Συνεπώς, συνάδελφοι, αν θέλετε να σας ακούσει ο συνάδελφος Ταραντ, προτείνω να είσαστε σύντομοι και θα συγχωρέσετε τον κύριο Ταράντ ο οποίος θα φύγει εκτός αν θέλετε κάτι να πείτε πριν ε, φύγετε κύριε Ταράντ παρακαλώ 11 λεπτά σε 11 λεπτά ωραία Τερμοντή ευχαριστώ πολύ πρόεδρε και εντάξει 11 λεπτά θα είμαι σύντομη πρώτον για τα σχόλια που έκαναν ε, και άλλοι. Και εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλή έκθεση αυτή. Τα σημεία που αναφέρει, η σαφήνεια, όλα αυτά είναι θετικά. Δύο ζητήματα. Το ένα είναι πληθωρισμός. Όπως είπε και ο Ζαμπόλ, ποιος είναι τελικά ο πληθωρισμός. Και δεύτερον, για να περιοριστούμε, έχουμε ε, τακτικές και έκτακτες δαπάνες η εμπειρία λέει ότι πάντα έχουμε έκτακτες δαπάνες. Οπότε ίσως να πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη μας από την αρχή, αντί κάθε χρόνο να μιλάμε για έκτακτες δαπάνες. Αυτό ήταν το πρώτο μου σημείο. Δεύτερο, ε, βάση επιδόσεων. Αν θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτή την αρχή, τότε χρειαζόμαστε πληροφορίες και διαφάνεια για να μπορούμε να τηρήσουμε αυτή την αρχή. Κυρίως όπως ακούσαμε όσον αφορά την ασφάλεια και τα κτίρια. Και κάποια άλλα ζητήματα λιγότερο ίσως σημαντικά. Ανταλαμβάνομαι αυτά που λέτε στην παράγραφο 20 ως εξής. Λέτε ότι συμμερίζεστε τις ανησυχίες ότι μερικοί θέλουν απλώς στατιστικά δεδομένα χωρίς να υπάρχει η σουσία από πίσω και ότι εσείς θέλετε περισσότερο ποιοτική εκτίμηση παρά ποσοτική. Και στην παράγραφο 21 θα ήθελα να προσθέσω κάτι το οποίο έχει ξανακουστεί, που είναι η δυνατότητα να έχουμε ανεξάρτητο έλεγχο για να κοστίζει λιγότερα όσον αφορά την γραμματιακή υποστήριξη, τα επιδόματα γραμματιακής υποστήριξης. Ευχαριστούμε κύριε Γανίζα ζαβάλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όσον αφορά την έκθεση του κυρίου Τάραν, λίγα πράγματα έχω να πω, γιατί οι σοσιαλιστές συμφωνούμε με τις προτάσεις που αναφέρονται στην έκθεση αυτή. Θέλω να επικεντρωθώ λοιπόν περισσότερο σε ερωτήσεις προς το Γενικό Γραμματέα, μια που τον έχουμε εδώ. Πρώτα ένα γενικό σχόλιο όμως. Πώς παρουσιάζεται ο προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί κάθε χρόνο βλέπουμε ότι έχουμε έναν προπολογισμό με έκτακτες ανάγκες. Και αυτές οι έκτακτες ανάγκες τον επόμενο χρόνο έχουν συμπεριληφθεί στον προπολογισμό. Δηλαδή βλέπουμε αιτιολογήσεις για περισσότερες δαπάνες και ποτέ δεν βλέπουμε να λέει επενδύσαμε αυτά για την προηγούμενη χρονιά, οπότε αυτή τη χρονιά δεν χρειάζεται να τα προβλέψουμε. Να προβλέψουμε δηλαδή τον προπολογισμό του έτους νη ε, με το προηγούμενο, ε, δεν θα έπρεπε να βλέπουμε αύξηση, ποτέ όμως δεν το διαπιστώνουμε αυτό. Ποτέ δεν μειώνεται κανένα απολύτως τμήμα. Όπως έλεγε και ο κύριος Λεανό, χρειαζόμαστε περισσότερη σαφήνεια το πού πάνε τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γι' αυτό θα έπρεπε να έχουμε διαφοροποιημένο προπολογισμό ανάμεσα με το αν μιλάμε για τρέχουσε δαπάνε ή επενδύσει. Γιατί οι τρέχουσε σαφώ και είναι σταθερέ, ενώ οι επενδύσει είναι πιο στιγμίε και έτσι θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε καλύτερα τα πράγματα. Και έρχομαι τώρα στην ασφάλεια και το σχεδιασμό τη. Ακούσαμε ότι δεν είναι καλύτερη στιγμή όταν είμαστε στις webstream να συζητήσουμε την κτηριακή πολιτική υπάρχουν έγγραφα τα οποία είναι απόρριτα, αλλά δεν έχουμε πληροφορίες για τις αποφάσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Εμείς είμαστε ε, σκέλος του προϋπολογισμού, συνεπώς πρέπει να έχουμε πληροφορίες για να μπορούμε να αποφασίσουμε πού θα επενδύσουμε. Χρειάζεται εδώ ισορροπία, γιατί άλλο είναι να μην έχουμε δημόσια όλα τα έγγραφα και άλλο είναι να έχουμε ελάχιστες πληροφορίες και ακόμα χειρότερα να έχουμε απλώς ένα κατάλογο θεμάτων που θα εξεταστούν φέτος και του χρόνου όσον αφορά την ασφάλεια. Δεν πιστεύω ότι θα αμφισβητήσει κανείς ή θα θέσει σε κίνδυνο τις δαπάνες ή θα αμφισβητήσει τις δαπάνες για την ασφάλεια. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να δούμε γενικότερα ώστε να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στις δαπάνες και την πραγματική απειλή. Συνεπώς το πρώτο είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίε. Και αυτό ισχύει και για τον σχεδιασμό των ε, κτηρίων μας μακροπρόθεσμα. Υπάρχουν πολλά σχέδια επιτάπητος. Και με το κτίριο PHS, το Poland Pack, τι θα το κάνουμε, μικρές αλλαγές, μεγάλη βελτίωση. Χρειαζόμαστε και πάλι λέω αρκετέ πληροφορίε για να μπορούμε να εκτιμήσουμε το κόστος και την αποτελεσματικότητα των σχεδίων που βρίσκονται μπροστά μας προς εκτίμηση. Έπειτα έρχομαι στο κεφάλαιο για τα 14 επιπλέον εκατομμύρια για να βοηθηθεί ο Ευρωβουλευτής στο έργο του. Και πάλι πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα βελτιωθεί με αυτό το Empowering Members Mandate όπως ονομάζεται με 14 επιπλέον εκατομμύρια ευρώ. Και θέλω να ξέρω γιατί το τμήμα εκείνο το οποίο έχει να κάνει με περισσότερους βοηθούς αυξάνεται. Πέρα από τον προϋπολογισμό κατά 1,7 και για τις υπηρεσίε έρευνας, τους εμπειρογνώμονες που κάνουν τις έρευνες αυτές. Εδώ στην Επιτροπή μας το είδαμε ότι την προηγούμενη φορά για την μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού πλαισίου είχαμε τρεις διαφορετικές έρευνες. Υπήρχε επικάλυψη. Γιατί δεν υπάρχει επικάλυψη. Και εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε τι υπηρεσίες υπήρχαν ήδη, το EPRS και τι χρειαζόμαστε. Επίσης θέλω να ξέρω πώς έχει κατάσταση όσον αφορά τους διερμηνείς, γιατί πέρυσι το ξανασυζητήσαμε. Είπαμε ότι υπήρχε ένα νέο σχέδιο εργασίας, συνθήκες εργασίας για τους διερμηνείς, που ήταν επίμαχο υπήρξαν προβλήματα στην υπηρεσία διερμηνίας. Γνωρίζουμε ότι για πολλούς και διάφορους λόγους υπήρχαν καμπύρες που χρειαστηκε να κλείσουν, δεν διασφαλίστηκε η πολυγλωσία, οπότε εγώ θέλω να γνωρίζω τώρα ποιες είναι οι προτάσεις που έχει υπόψη του και έχει υποβάλει ο Γενικός Γραμματέας. Ναι, μια μισή ώρα, ξέρω, έχει ήδη περάσει ο χρόνος, δεν φτάνει όμως για να μπορεί κανείς να αποφασίσει, ξέροντας τι κάνει, χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κυρία... Για την Μάκη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ακόμη πιστεύω ότι θα ήταν ε, καλή ιδέα να έχουμε περισσότερη ενημέρωση όσον αφορά την ε, ασφάλεια, την ανακαίνιση των κτίριων και την πολιτική των ε, ακινήτων γενικότερα. τον έχουμε ένα καταβογωπή ποσό ε, για κανένα από αυτούς τους τομείς. Θα πρέπει οι παλιοί να γνωρίζουν ακριβώς πότε προϋπολογισμός υπάρχει για τα οικοδομήματα. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι όσον αφορά ασφάλεια, τα ακίνητα και την ανακαίνιση. Επίσης, δύο λόγια θα πρέπει να αναφερθούν για την ενιαία μία μοναδική έδρα και το Στρασβούργο. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Πριν μας εγκαταλείψει για τη χώρα του, όπου θα πάει να ερωτάσει το 98 χρόνια της δημοκρατίας στην Εστονία, θα σας δώσουμε το λόγο κύριε Ισηγητά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όχι, δεν είναι γιατί δεν σέβομαι την διαδικασία επί του προπολογισμού, αλλά η μέρα ανεξαρτησίας ε, είναι πάρα πολύ σημαντική μέρα. Είναι ευρωπαϊκή μέρα για μας και λαμβάνω υπόψη όλες αυτές τις ε, προτάσεις από όσους έλαβαν τον λόγο στη συζήτηση και οι οποίοι ε, υπέβαλαν κάποιες παρατηρήσεις, κάποια σχόλια και πάλι εγώ προσπαθώ να σας πείσω για το ότι κατά τη γνώμη μου ο Γενικός Γραμματέας ε, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά με τις πληροφορίες που μας έδωσε. Το θέμα είναι βέβαια το ότι πολλές φορές έχουμε κάποιες πολύ στοχευμένες συγκεκριμένες ερωτήσεις οπότε ελπίζω τελικά να τα πάμε καλά, να τα καταφέρουμε. Ξέρουμε πάντως ότι εδώ έχουμε διαφορετικά κόμματα, διαφορετικές πολιτικές ομάδες και πρόκειται τελικά να υποβληθούν τροπολογίες τις οποίες και θα επεξεργαστούμε δεν θα μπορούσα τώρα στο σχέδιο του, κειμένου να καλύψω όλα τα επιχειρήματα. Προσπάθησα να βρω τη μέση εδώ κατά κάποιο τρόπο και επίσης όπως θα παρατηρήσατε έχουμε αυτόν τον ε, υπολογισμό, αυτό τον τύπο υπολογισμού του πληθωρισμού που θα πρέπει να το ξανακοιτάξουμε. Εγώ αντιλαμβάνομαι επίσης ότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ε, θα πρέπει να κατεβάσουμε το κείμενο στην Ολομέλεια του Απριλίου. Αυτά επομένω. και συμπαθάτε μου θα πρέπει να φύγω από την σημαντική μας ε, συνάντηση. Ο πρόεδρος. Μαζί σας θα είμαστε αύριο, να ξέρετε κύριε Ταράντ. Οι διερμηνείς θα πρέπει να φύγουν στις 16 και 45. Συνεπώς όσοι πάρουν το λόγο, παρακαλώ να είναι σύντομοι. Παρακαλώ, κύριος Μακάου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα επικεντρωθώ σε δύο στοιχεία κλειδί. Δεν θα μακρηγορήσω, πολλά θα μπορούσε κανείς να πει, αλλά να, σαν παράδειγμα. Όταν ετοιμάσαμε τον προπολογισμό του 2015, είχαμε σκεφτεί ότι τακτικές ε, δαπάνες έπρεπε να αυξηθούν κατά 1,7%. Και αν δείτε ότι το τωρινό ε, πληθωρισμό ήταν 0,5% το 2015 έτσι στο Λουξεμβούργο, 0,6% στη Γαλλία κτλ. Έχουμε λάβει υπόψη μας όλες τις τιμές αγαθών βάσει δικτών, αλλά οι δείκτες που έχουμε χρησιμοποιήσει για την προσαρμογή πολλές φορές δεν ήταν ρεαλιστικοί. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τους πραγματικούς δείκτες. Αλλιώς σε 50 χρόνια από τώρα θα υπάρχει μια πλήρη στρέβλωση των ε, ποσών. Θα ήταν καλό λοιπόν να Υπάρχει προπολογισμό κάθε πέντε χρόνια που να βασίζεται στις τρέχουσες ε, τιμές και δαπάνες. Και μετά ανάλογα να προσαρμόζεται αν χρειάζεται. Δεύτερον, κύριε Γενικέ Γραμματέα, εγκρίναμε τις δαπάνες για την ασφάλεια για το 2015 και οι δαπάνες αυτές είπαμε ότι θα είναι αναγκαίες και για το 2016 και για το 2017. Ναι, πρέπει όμως να έχουμε ένα συνολικό σχέδιο, να γνωρίζουμε ποιο ακριβώς είναι το κόστος και τι περιλαμβάνει. Το 2016 έχουμε 15 εκατομμύρια, το 2017 θα είναι 30 εκατομμύρια και βρισκόμαστε στο σκοτάδι. Δεν είναι καλός τρόπος ε, εκπόνησης του προπολογισμού να έχουμε ένα συνολικό σχέδιο που να ξέρουμε τι περιλαμβάνει και τι θέλουμε να πετύχουμε με αυτό. Και έχουμε στο τελευταίο μου. Έχουμε γραπτές ερωτήσεις που έχουμε ετοιμάσει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 60 από, απαντήθηκαν από την Επιτροπή. Μιλήσαμε για μείωση των δαπανών όμως εγώ νομίζω ότι πρέπει αυτό να αντικατοπτρίσετε στον νέο προπολογισμό και να χρησιμοποιούμε τους ήδη υπάρχοντες πόρους, το προσωπικό δηλαδή, χωρίς να προσλαμβάνουμε καινούριους. Ο κύριος Γιώτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έργο του. Εγώ θέλω ε, να αναφέρω μόνο σε δύο θέματα τα οποία δεν ε, σχολιάστηκαν γιατί κατά τα λοιπά ε, καλύπτομαι από τους συναδέλφους της ομάδας μου ή των άλλων συναδέλφων που συμφωνώ μαζί τους. Θα ε, σας πω το εξής. Εδώ στην Επιτροπή μας όταν έχουμε συνεδρίαση ε, έχουμε πιο πολλές ε, συνεδριάσει ε, των υπευθύνων για τα κτίρια παρά αυτές που κάνουμε εμείς γιατί μιλούμε τώρα για νούμερα για κάποια στοιχεία για κάποια έργα τα οποία αφορούν τις ε, αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου σε όλο τον κόσμο, τα γραφεία του Κοινοβουλίου. Άρα θα πρέπει να διαθέσουμε περισσότερο χρόνο αντί για αυτά στα πιο πολιτικά ζητήματα. Επίσης, να σας πω κάποιες άλλες σκέψεις μου. Θεωρώ ότι προκαλεί αρκετή έπληξη αυτό το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε φορά που μιλούμε για τη διαχείριση των ε, ακινήτων των θεσμικών οργάνων και του Κοινοβουλίου το πώς έχουν παλιώσει τα κτίρια που είναι 25-30 ετών και σας ε, υπενθυμίζω ότι το κτίριο του Γαλλικού Κοινοβουλίου φτιάχνει 1722 και 1650 στην Ιταλία και το 1992 το πιο παλιό, το Βρετανικό και το Αγγλικό Κοινοβούλιο. Οπότε μιλούμε για, τώρα για κτίρια ε, παλιά. Ε, αυτό νομίζω ότι είναι εσφαλμένο. Είναι θέμα της συνήθους διαχείρισης των κτίριων μας. Αυτό θα πρέπει να λέμε. Και να μην έχουμε νερό στο μήλο των ευρωσκεπτικιστών ε, με τα έξοδα αυτά. Τώρα κάτι άλλο. Για πέστε μου. Πώς είπατε. Ναι, ναι, ναι, κλείνω, κλείνω πρόεδρε. ακριβώς τι γίνεται με το κοινοβούλιο πού θα βρούμε κάποια στοιχεία για το στόχο ε, για κατά πόσο είναι στόχος δηλαδή το κοινοβούλιο είναι θέμα άμεσο ή ασφάλεια άρα θα πρέπει να κάνουμε κάτι τώρα άμεσα και να μην κάνουμε κάτι μέσω του προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου. Να είπαμε να έχουμε εσωτερικούς ε, ε, οδηγούς. Αν είναι όμως θέμα ασφάλειας θα πρέπει κανείς να λάβει μέτρα άμεσα και να μην περιμένει την έγκριση ενός προϋπολογισμού. Αν πρόκειται για γενικό, γενικευμένο κίνδυνο, τότε αυτό θα πρέπει να κάνουμε, να λάβουμε μέτρα. Και βέβαια, αν είναι θέμα δικαιωμάτων των εργαζομένων θα πρέπει να τα σεβαστούμε και να έρθουμε σε επαφή με τους κατάλληλους φορείς. Αυτές είναι οι σκέψεις που θέλω να σας πω και σας ευχαριστώ και τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές για τη δουλειά τους. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Δόσκη. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Κύριε Γενική Γραμματέα. Και κύριε Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είσαστε και ο αγαπημένο μου Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνεισηγητέ, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ όλους για την υπέροχη αυτή έκθεση. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά τα οποία έχουν ήδη τεθεί. Νομίζω ότι σένα πρέπει να σταθούμε. Το σημείο 28 ο εισηγητή εκφράσει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την μετάφραση και τη διερμηνία. Το έχουμε συζητήσει αυτό με τον κύριο Βέλε και έχουμε πει τι πρέπει να κάνουμε. Όταν λέτε ότι υπάρχει πρόοδος, τι ακριβώς εννοείται. Σήμερα το πρωί είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού και υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην ποσότητα και την ποιότητα όταν μιλάμε για τη διερμηνία. Πιστεύω ότι η ποιότητα είναι αυτή που πρέπει να κυριαρχεί και όχι τα νούμερα όσον αφορά το πόσοι διερμηνείς ε, κάναν τι και πόσες ώρες απασχολεί το καθένα τους. Η ποιότητα λοιπόν είναι πιο σημαντικό. Ευχαριστώ. Κύριε Σωστοφόρου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γραμματέα, ε, πιστεύω ότι αυτή τη συζήτηση την επαναλάβαμε και πέρσι. Έγινε εξαντλητική συζήτηση για τον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δυστυχώ επαναλαμβανόμεθα. Και πιστεύω έγινε και από τον κύριο Ντεπρέ εξαιρετική δουλειά πέρσι και φέτο από τον κύριο Ντάρα. Και όλοι λέμε και ανησυχούμε ότι, ξέρετε, με τη συζήτηση για τον προπολογισμό τάχατε σε ευαισθητοποιούνται οι ευρωσκεπτικιστέ, δημιουργείται ζημιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα αφού εμεί ήδη αναδεικνύουμε αυτά τα ζητήματα. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτοπυροβολείται. Ο προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι το 1% ολόκληρου του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ασχολούμεθα με το 99% που εκεί υπάρχουν πολλέ δυνατότητε, να μην πω σπατάλε δυνατότητε να εξοικονομήσουμε πολύ περισσότερα χρήματα. Επικεντρωνόμαστε στο 1% πολλέ φορέ με λεπτομέρειε και με τρόπο για να αναδειχθούμε ότι τάχατε εμεί είμαστε αυτοί οι οποίοι υπερασπιζόμαστε τα κονδύλια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στο τέλο αυτό που θυματοποιείται είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ θεωρώ ότι με το 1% του προπολογισμού που έχουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με ένα ισχυρό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελέγχουμε καλύτερα τι δαπάνε του άλλου 99% αλλά και τι δικέ μα και έχουμε τεράστιε εξοικονομήσει. Εάν κάθε χρόνο ερχόμαστε και αποδυναμώνουμε την ισχύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο τέλο είναι τεράστια ζημιά στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση που κάνουμε και εκεί είναι που ενισχύουμε του ευρωσκεπτικιστέ Δημιουργώντα έναν αδύνατο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα άλλο πολύ σημαντικό για μένα είναι ότι και επειδή γίνονται τεράστιες αναφορές για το τι δίνεται για του ευρωβουλευτές μα να σας πω κάτι και δεν γίνεται ποτέ καμιά αναφορά για κανέναν άλλο σώμα όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωση, απλώς να αναφέρω σε δεικτικό για να δείτε τι παραπληροφόρηση γίνεται ο μισθός του ευρωβουλευτή είναι το 33% του μισθού του δικαστή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ποτέ δεν αναφέρθηκε αυτό το πράγμα και ποτέ δεν ασχολήθηκε κανένα με του μισθού κάποιον άλλο. Εμεί που λαμβάνουν το 33 ασχολούμεθα εμεί ήδη και τον αδεικνύουμε, ενώ για του άλλου για χάρη τη δημοσιότητα ουδή ασχολείται. Εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήρθε και αύξησε τι πράσινε εβδομάδε, που θέλω να ξέρω από το Ευρωκοινοβούλιο και από τον κύριο Γραμματέα τι εξοικονομήσει είχαμε που ήταν σωστή ενέργεια και μπορούν να αυξηθούν ακόμα περισσότερο γιατί και ουσιαστικά προσφέρουν γιατί δίνουν τη δυνατότητα στους ευρωβουλευτέ να είναι στι χώρε του, γιατί είναι πολιτικά δραστήρια άτομα και δεν είναι απομονωμένα στο Ευρωκοινοβούλιο, ενώ κάναμε αυτήν την τεράστια πραγματικά εξοικονόμηση και νοικοκύρεμα, όχι μόνο δεν το αναφέρουμε, ξαναρχίζουμε από την αρχή τα ίδια και τα ίδια. Θα ήμουν και εγώ πολύ άρεστος, ιδιαίτερα τώρα που μεταδίδεται, να πω να κοπούν όλα θα ήμουν πολύ αρεστό να πω ότι να υπάρχει ένα Ευρωκοινοβούλιο που να είναι στο επίπεδο του, εργαζομε... του μέσου εργαζομένου στι Βρυξέλλε. Και με αυτόν τον τρόπο τελειώνω κύριε Πρόεδρε με μια φράση. Αυτό που πρέπει να μα απασχολήσει είναι η ποιότητα του έργου. Και η ποιότητα του έργου αναδεικνύεται και με τη μείωση τη γραφειοκρατία και κανένα δεν αναφέρθηκε. Αυξήθηκε η γραφειοκρατία. Και θα πω ένα σημείο που είναι σημαντικό και πρέπει να το επιλεξεί ο γραμματέα. Πολύ ορθά ο κύριο Ντεπρέ περιέρισε τι ερωτήσει. Έβαλε τέσσερι ερωτήσει επίγουσες. Μακάρι να καταριόντουσαν και αυτέ, να μην υπήρχαν. Κάνει την επίγουσα ερώτηση και αποφασίζει άλλον όργανο να είναι επίγον. Και επανέρχεται πίσω η ερώτηση και σου λένε ότι δεν είναι επίγουσα ερώτηση γιατί έτσι κρίναμε και πρέπει να την ξανακάνει. Αυτό το πράγμα είναι γραφειοκρατία, είναι κόστο, είναι επιβάρηση. Θέλουμε να μειωθεί η γραφειοκρατία και πιστεύω συμφωνώ με όλου του συναδέλφου και όσα είπα δεν έχω αντιπαράθεση με κανένα να επικεντρωθούμε περισσότερο στη μείωση τη γραφειοκρατία που θα περιορίσουμε δαπάνε και θα αναδείξουμε και καλύτερα τον ρόλο του Ευρωβουλευτή. Ευχαριστούμε. Τελευταίος. Είναι αλήθεια ότι βαραίνει λίγο ο προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με το συνολικό προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτόν μπορούμε εμεί να επηρεάσουμε πολύ. Και όλα εξαρτώνται από το πόσο εμείς θα πειθαρχήσουμε και πόσο εμείς θα ελέγξουμε λεπτομέρω. Δεν υπάρχει. Μιλάμε για την καλύτερη νομοθέτηση. Όταν νομοθετούμε λιγότερο, Πώ γίνεται να αυξάνονται οι δαπάνε κατά 3,9%. Ακούσαμε διάφορα επιχειρήματα, αλλά όταν μιλάμε για περιορισμό των δημοσίων δαπανών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου, πολύ προσοχή. Θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Πέρυσι, με έκπληξη, μάθαμε την αύξηση των μισθών, ενώ ο προπολογισμό είχε φτιαχτεί βάσει άλλων υπολογισμών. Πήρατε τα μέτρα σας ώστε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία να δίνει στατιστικούς δείχτες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να έχουμε στοιχεία πολύ νωρίτερα και να μην υποστούμε και πάλι σοκ που ήταν σοκ όταν τελευταία στιγμή μάθαμε για αυτή την αύξηση. Έπειτα, εγώ θέλω ο προπολογισμό να είναι κανονικός. Να είναι ετήσιος. Για το 2016 είπαμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνική των προεδρικών μεταφορών. Θα ήθελα να μας επιβεβαιώσετε ότι τηρούμε το, την, το ενάψιο του προπολογισμού, ότι δηλαδή είναι ετήσιος. Και να μας πείτε γιατί κάποιες μεταφορές, κάποια εμβάσματα είναι προεδρικά και κάποια άλλα όχι. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πέρα. Θα επιχειρήσω τουλάχιστον θεματολογικά να δώσω απαντήσεις. Κάποιοι τοποθετήθηκαν στο ίδιο θέμα και θα προσπαθήσω να αποφύγω τις υπερβολικές επανάσεις. Ε, και πρέπει να διαχειριστούμε και το χρόνο. Για τον πληθωρισμό η αξιολόγηση, η εκτίμηση του πληθωρισμού γίνεται επί τη βάση μιας πρότασης επιτροπής, μιας εκτίμησης επιτροπής, πάνω στην οποία όλοι στηριζόμαστε και εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που αποτελεί την βάση εκκίνησης για τον υπολογισμό του πληθωρισμού. Δεν είναι δηλαδή τα νούμερα δικά μας και αυθαίρετα, είναι νούμερα τα οποία χρησιμοποιούμε για όλους τους προϋπολογισμούς. Δεύτερον, ανακαίνιση στα καινούρια κτίρια κάθε 25-30 το πολύ έτη γίνεται ανακαίνιση. Πρέπει να γίνει πρόβλεψη για ανακαίνιση. Στα πιο γυραιά κτίρια επίσης ισχύει το ίδιο. Δόθη το παράδειγμα του Westminster. Το Westminster καθυστέρησε πολύ την ανακαίνιση του για πολλά χρόνια γιατί προτιμούν οι βουλευτές της Βουλής των Κοινοτήτων να συνεδριάζουν στο Westminster Palace και σε κάποιο ανώνυμο κτηριακό συγκρότημα. Και τώρα από ό,τι μαθαίνω θα φτάσει στα δισεκατομμύρια, ίσως και έξι δισεκατομμύρια λίρες το κόστος γιατί θα χρειαστεί εκβάθρον ανακαίνιση. Όταν περάσει δηλαδή ένα συγκεκριμένο χρονικό ε, διάστημα, όριο στο οποίο απαιτείται να γίνει η ανακαίνιση, τότε γίνεται σημαντικά πιο ακριβή το κοινοβούλιο. Δεν έχει χτίσει κανένα κτίριο μόνο του. Το ΚΑΤ έχει οικοδομηθεί ως συνεδριακό κέντρο από, έναν, από μια σύμπραξη ιδιωτική εταιριών από την οποία αγόρασε το κτίριο το κοινοβούλιο. Και αναλόγως κινούμαστε και για τους ποντικούς που ίσως να έχουν πάρει θρηλυκές πλέον διαστάσεις, υπάρχουν ε, απαντήσεις. Υπάρχει ένα ηλεκτρικό σύστημα για το οποίο Φερρυπίν δεν προβλέπονται καν ανταλλακτικά. Εάν τυχόν ε, σταματήσει να λειτουργεί θα χρειαστεί ίσως και να κλείσει κτίριο γιατί είναι παλιές οι εγκαταστάσεις. Όλα αυτά πρέπει να τα προβλέψουμε και να προχωρήσουμε στην ανακαίνιση του κτίριου. Και άρα το ζήτημα είναι μάλλον το πώς θέλουμε να κάνουμε την ανακαίνιση όχι το αν θα την κάνουμε. Κάνουμε μια απλή αντικατάσταση των ε, τεχνολογικών υποδομών ή ανοίγουμε ένα πιο φιλόδοξο έργο τεχνολογικό και ενεργειακό ή και δίνουμε επιπλέον δυνατότητες για το μέλλον στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κτίρια του, γιατί ε, το έθιξα νωρίτερα. Εάν αυξηθούν τα κράτη-μέλη και άρα και οι γλώσσες, θα, θα κληθούμε να δώσουμε απαντήσεις στο εάν συνεχίζουμε την πολυγνωσία όπως έχει έως τώρα. Και αν είναι αυτή η απόφαση θα πρέπει να προβλέψουμε τις σχετικές εγκαταστάσεις ε, συνεδριάσεων, αίθουσε συνεδριάσεων και το καθεξής με καμπίνες ώστε να καλύπτεται από τη διερμηνία η πολυγλωσία η μία ή η άλλη επιλογή είναι φυσικά πολιτικές αποφάσεις. Η οδηγή. Ξέρετε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή εξωτερική υπηρεσία οδηγών που γεγονός το οποίο οδηγεί σε κάποιες δυσκολίες. Καταρχάς το θέμα της ασφάλειας, της ασφάλειας που πρέπει να συζητήσουμε ξεκάθαρα και ανοιχτά, αλλά και πέραν αυτού το θέμα των κοινωνικών προδιαγραφών, το θέμα του σωστού μισθού, ε, τις αποζημίωσεις για υπηρεωρίες, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ίσως μπορούμε εμείς καλύτερα να καλύψουμε εσωτερικά από το να έχουμε μια εξωτερική υπηρεσία που αλλάζει καθημερινά προσωπικό ε, οδηγών και έτσι δεν ξέρουμε ποιος έρχεται στα αυτοκίνητα. Επίσης, αν υπάρχει δυνατότητα για εις βάθος συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών και την ε, Οικονομική και Πολιτική Επιτροπή, ετέθη το ερώτημα. Έχουμε μια πολύ καλή εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια. 60 οι υπάλληλοι της, ε, των Επιτροπών ήρθαν στο Κοινοβούλιο με πολύ καλά, καλή δουλειά, πολύ ποιοτική δουλειά χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση για τον φορολογούμενο. Δηλαδή μπορέσαμε να ενισχύσουμε την επιστημονική μας υπηρεσία εμείς, η δε ε, δύο αυτές συμβουλευτικές επιτροπές για πρώτη φορά έχουν στα θέσή τους τις υπηρεσίες μιας επιστημονικής ε, υπηρεσίας. Και έτσι υπάρχει αυτή η συνεργασία, υπάρχει ενισχυμένη συνεργασία και ως προς την πληροφορική και σε περίπτωση ε, ενισχυμένων αναγκών και για τη μετάφραση και για την ασφάλεια. Υπάρχει δηλαδή στον τομέα αυτών συνεργασία η οποία ασφαλώς μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω, να εμπαθυνθεί. Για τις γλώσσες. Το Κοινοβούλιο επιμένει να εργαζόμαστε σε όλες τις γλώσσες. 24 σήμερα, 25 ίσως αύριο, ίσως και 30 μεσοπρόθεσμα εφόσον πρόκειται για ένα θεμελιώδες δημοκρατικό δικαίωμα. Εάν όμως θέλουμε να το εγγυηθούμε αυτό για το μέλλον, πρέπει να οργανώσουμε αποτελεσματικά τις γλωσσικές υπηρεσίες. Ο συνδυασμός της διευρύνσεως της γλωσσικής κάλυψης και της μη αποτελεσματικής οργάνωσης είναι κατά την δική μου θεώρηση καταστροφικός. Γι' αυτό και έλαβε μια σειρά αποφάσεων πέρσι το Κοινοβούλιο προκειμένου να οργανώσει πιο οικονομικά αυτές τις υπηρεσίες, δηλαδή καλύτερο προγραμματισμό των συνεδριάσεων των επιτροπών, αποφυγή των νυχτερινών συνεδριάσεων για να, γιατί μετά δεν θα μπορούν την επόμενη μέρα να εργαστούν οι διερμηνείς, καλύτερη αξιοποίηση των γλωσσικών υπηρεσιών στα ταξίδια στο εξωτερικό του Κοινοβουλίου, στις αντιπροσωπείες, αλλά πολλά ακόμα μπορούμε να κάνουμε και οφείλουμε να πράξουμε τα επόμενα χρόνια Άρα ζητήματα της αποτελεσματικότητας ε, είναι ζητήματα τα οποία δεν θεωρούμε δευτερεύοντα αλλά κέρια σημασίας προκειμένου με τις νέες αυτές συνθήκες προκύπτουν να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την παροχή της πολυγλωσσίας ως υπηρεσίας με την ποιότητα ασφαλώς. Γι' αυτό και συνομιλούμε και με τους διερμηνείς εντατικά. Το έχω πράξει εγώ προσωπικό στις αρχές του χρόνου και θα συνεχίσω τον διάλογο. Για το θέμα των μίνι παρλαμεντάριου το Προεδρείο αποφάσισε να εγκαθιδρύσει δύο Παρλαμεντάριου είναι Παρλαμεντάριου, ένα στο Στρασβούργο, όπου και στο Στρασβούργο έχουμε πάνω από 100.000 επισκέπτες το χρόνο, έξω από τις εβδομάδες της Ολομέλειας επίσης. Μάλιστα αυτό θα μας είναι σχετικά οικονομικό σαν λύση, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία έτσι να προσφέρουμε ε, την ενημέρωση στον πολίτη και έξω από τις συνεδριάσεις της Ολομέλειας. Έχει εγκριθεί Επίσης η πρόταση για ένα μίνι παρλαμεντάριο στο Περβερολίνο εγκρίθηκε από το Προεδρείο. Είναι πολύ ε, ε, εύστοχη επιλογή της θέσεώς του κοντά στην πύλη του Βραδεμβούργου με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και άρα πιστεύουμε ότι με σχετικά περιορισμένο κόστος ε, μπορούμε να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες χωρίς να χρειάζεται να έρθουν μέχρι τις Βρυξέλλες ή το Στρασβούργο. Εάν λοιπόν στεφθεί με επιτυχία αυτό το εγχείρημα μπορούμε ασφαλώς να αναλογιστούμε αν υπάρχουν δυνατότητες και κατάλληλες τοποθεσίες για αντίστοιχες άλλες εγκαταστάσεις. Πάντως Προς το παρόν διαπιστώνουμε, ε, πρέπει να παραμένουμε στη διαπίστωση του αν είναι επιτυχημένο το εγχείρημα ή όχι. Αυτό θα είναι το επόμενο βήμα, θα πρέπει να το αποφασίσει βέβαια το Προεδρείο. Εάν δεν είναι επιτυχημένη η πρόταση, θα πρέπει να αντληθούν τα σχετικά συμπεράσματα. Για τα μπαούλα που μεταφέρουν το ε, τα έγγραφα και εδώ έχουν γίνει πολλές προτάσεις. Η χρήση αυτών των μπαούλων θα μπορούσε να περιοριστεί πρώτον και αυτό το ανέφεραν αρκετοί βουλευτές, βουλευτές το κάνουμε στο δυνατόν περισσότερο στη διοίκηση, δηλαδή ενημερώνουμε λέγοντας ότι πρέπει να γίνεται χρήση ενός μπαούλου από περισσότερους ε, υπαλλήλους Κάποιοι μπορεί να μην χρειάζονται καν ε, τον μπαούλο ή να χρησιμοποιούνται πιο μικρών διαστάσεων μπαούλα. Προσπαθούμε όπως ε, και να, κάνουμε οικονομία στο τομέα αυτών. Για την ασφάλεια. Θα συνιστούσε βαρύτατη αμέλεια πιστεύω το να μην αντιδράσουμε αναλόγως της υφισταμένης κατάστασης σε σχέση με την ασφάλεια εγώ προσωπικό και πιστεύω και το Προεδρείο, το είδε και ο Πρόεδρο ο ίδιο, δεν είμαι διατεθειμένη να λάβω αυτή την ευθύνη. Και γι' αυτό και διατυπώνουμε αυτέ τι προτάσει. Είναι γνωστό εντωμεταξύ πώ έχει αλλάξει η κατάσταση σχετική με την απειλή. Όλε οι είσοδοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες ασφαλείας ή ε, διακινδύνευσης αντίστοιχα ασφαλεία η διακινδύνευση, αντιστοιχα και όπω ειπαμε εγινε η προσαρμογη τη εισόδου από την πλευρά πλατείας Λουξεμβούργου στις Βρυξέλλες. Αυτές είναι οι νέες εξελίξεις και κατά τη διάρκεια του 2016 και του 2017 θα γίνουν οι εγκαταστάσεις στις λοιπές εισόδους. Εδώ προτείνουμε τα κονδύλια τα αντίστοιχα για το 2017. Καθώ όμω θα συνεχιστεί αυτή η δουλειά και ο προγραμματισμό κατά τη διάρκεια του 2016, θα αντλήσουμε κονδύλια από λιγότερο επίγοντα καθήκοντα, προκειμένου να εξοπλίσουμε και τις, λιπότε, τις λιγότερο σημαντικές εισόδους ε, του κτηρίου των Βρυξελών με ε, επενδυ... έτσι ώστε να μπορούν να επενδυθούν και να φτάσουν ε, στο ύψος των αναγκών. Ενίσχυση των βουλευτών στα γραφεία τους στις χώρες μέλη, στις πατρίδες τους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια παρεξήγηση εδώ. Έχουμε 14 εκατομμύρια όχι επιπλέον όμως κονδύλια, είναι ε, διαθέσιμα κονδύλια σε σχέση με το προηγούμενο έτος που θα αξιοποιηθούν ιδιαίτερως για την ενίσχυση της ε, των πληροφορικής και των υποδομών και θα γίνει προσαρμογή έτσι ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν όχι μόνο τις έδρες του Στρασβούργου και των Βρυξελών αλλά και στα γραφεία των βουλευτών στις χώρες τους μπορούν να αξιοποιηθούν ε, εγκαταστάσεις ε, βίντεο διασκέψεως δεν θα πρόκειται δηλαδή για νέες εγκαταστάσεις τεχνικές ή ε, νέα κονδύλια, αλλά και χωρίς αλλαγή για το τι είδου ε, πρόγραμμα θα χρησιμοποιείται κανείς στο υπολογιστή του στο Στρασβούργο της Βρυξέλλες ή και στο γραφείο του στις, στην πατρίδα του μπορεί να έχει αυτή την επικοινωνία. Μια ελαφρά προσαρμογή του προϋπολογισμού έχει να κάνει με την δυσκολία σε σχέση με τη ζήτηση και γι' αυτό είχαμε μια ελαφρά προσαρμογή καθώς το Προεδρείο αποφάσισε να αλλάξει τους κανόνες για τους βοηθούς. Ουσιαστικό, ε, ουσιαστική συνέπεια της εκθέσεως για την εκτέλεση του προπολογισμού του 2015. Νέοι κανόνες λοιπόν και νέα κονδύλια που απορροφούνται σε επίπεδο Βρυξέλλες, το, Βρυξελών, τώρα και στις ε, έδρες των, στις χώρες ε, μέλη τέλο πάντων. Υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση λοιπόν για βουλευτές, για βοηθούς συγγνώμη, των βουλευτών και αντίστοιχα εγκαταστάσεις. Και δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς θα εξελιχθεί το σχετικό κόστος, γι' αυτό βρισκόμαστε όπως βλέπετε ε, σε θέση να με μόνο μία πολύ προσεκτική προσαρμογή του προϋπολογισμού. Το ζήτημα της έδρας δεν το αποφασίζει το Κοινοβούλιο, οπωσδήποτε όχι η διοίκησή του. Είναι κάτι το οποίο ορίζουν οι συνθήκες και ε, ως εκ τούτου και εμείς οφείλουμε και μόνο να το σεβαστούμε. Μισθή. Εμείς εδώ τηρούμε τις ε, προσεγγίσεις και επιλογές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει μία σχετική εξέλιξη με βάση τον τη Μάρινθο, τη Μάρινθο στα κρατη σε κάποια κράτη-μέλη συγκεκριμένη και ανάλογα προτείνει την αύξηση των μισθών. Ξέρετε ότι έχετε, έχει, ε, διαπράξει σφάλμα και προς τις δύο κατευθύνσεις, και προς την κατεύθυνση της μείωσης και προς την κατεύθυνση της αύξησης των μισθών ε, τα τελευταία χρόνια. Ο πρόεδρος Δεκόπτη. Αν μου επιτρέπετε, μας εξηγήσατε πέρσι ότι επειδή η Eurostat δεν ήταν σε θέση να δώσει στοιχεία τη στιγμή όπου καταρτιζόταν ο προϋπολογισμός, ε, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είχαμε αυτή την στρέβλωση στα στοιχεία. Και ως εκ τούτου, αναδρομικά από 1η Ιουλίου του 2015 δόθη η αύξηση. Αυτό καταγράφηκε ως δυσλειτουργία και κάποιο πρέπει να βρούμε μια λύση για να το αντιμετωπίσουμε. Ο Γενικός Γραμματέας, να σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής δεν υπάρχει χωριστή αξιολόγηση από το Κοινοβούλιο, από τη διοίκηση του Κοινοβουλίου της υπόθεσης των μισθών. Η Επιτροπή έχει μια βάση υπολογισμού και σε αυτήν προσαρμόζονται και υπολογίζουν όλα τα θεσμικά όργανα τους ε, προϋπολογισμούς για, τις, για τους μισθούς. Δεν μπορούμε δηλαδή εμείς να βασιστούμε σε διαφορετικές βάσεις υπολογισμού ή υποθέσεις εξελίξεων του τιμαρίθμου. Πώ είπαμε, προσαρμοζόμαστε στι προτάσει τη επιτροπή. Προ τη μία προς την άλλη κατεύθυνση, είτε προ τα άνω, είτε τα κάτω. Για τα εμβάσματα. Ε, βεβαίως και ακολουθούν το δημοσιονομικό κανονισμό. Είναι ξεκάθαρο το ποια είναι τα εμβάσματα τα οποία εγκρίνει η ίδια η Επιτροπή των Προπολογισμών. αλλά βεβαίω και ο πρόεδρος ε, του ε, Κοινοβουλίου μπορεί για πολύ πιο περιορισμένα ποσά και πολύ αυστηρά καθορισμένου τομεί να εγκρίνει μόνος του εμβάσματα. Είναι κάτι το οποίο ε, αξιοποίησε ως δυνατότητα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 1,8 δις ήταν ο συνολικός προϋπολογισμός και ήταν 2-3 ε, εκατομμύρια μόνο το ποσό των εμβασμάτων που ενέκρινε ο ίδιος ο πρόεδρος ε, του Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε πολύ και Γενική Γραμματέα. Ο κύριο Βίλαντ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ σύντομα. Θα πρότεινα την επόμενη φορά κομμάτι τη αδείας τη επιτροπή των προπολογισμών να γίνει και κλεισμένων των θυρών, ώστε να μπορούμε να συζητήσουμε πιο διεξοδικά και αναλυτικά τα θέματα της ασφάλειας. Πρώτο. Δεύτερο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κοστίζει 3,6 ευρώ στον κάθε πολίτη σε σχέση με τα εθνικά κοινοβούλια, γιατί είναι πολύ λιγότεροι κάτοικοι ίσως. Αλλά εάν συγκρίνουμε με το Αμερικανικό Κοινοβούλιο αντίστοιχα, αυτό κοστίζει 5 ευρώ στον κάθε πολίτη. Ένα τρίτο μάλιστα του κόστους εμείς το έχουμε λόγω της έδρας και των γλωσσικών υπηρεσιών. Λοιπόν, ως κοινοβούλιο είμαστε πολύ οικονομικό, φθηνό εντός εισαγωγικών κοινοβούλιο. Δεύτερον ή τρίτον, κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να μας απασχολήσει σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα το ζήτημα της ε, παρουσίασης του προϋπολογισμού. Γιατί έφυγε πολλές φορές το ζήτημα αυτό. Ίσως ήταν καλό να έχουμε μια διαφορετική παρουσίαση του προϋπολογισμού. Ίσως θα πρέπει να αλλάξουμε σύστημα παρουσίασης. Ίσως θα πρέπει να δείχνουμε και τους επιμέρους προϋπολογισμούς των επιτροπών. Τις ώρες εχμής όπου είναι πιο ακριβή η διερμηνείς από τις, άκρες θα έλεγα της ε, εργάσιμης εβδομάδας και αναλόγως να κάνουμε τους υπολογισμούς μας. Δεν νομίζω όμως κύριε Πρόεδρε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ε, μπορεί να εξεταστεί όταν είναι εν εξελίξει εργασίε ε, τη Επιτροπή. Α κάνουμε λοιπόν το Σεπτέμβριο που έχει κλείσει λίγο πολύ ο χρόνο μια ακρόαση για να δούμε τι είδου δομέ θέλουμε για τον προπολογισμό μα για τα επόμενα χρόνια, πώ μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάρτιση και την παρουσίαση του προπολογισμού. Ποσοτική προσέγγιση. Με κατέπληξε το γεγονό ότι κανεί δεν τοποθετήθηκε συγκεκριμένα σε αυτό. Έριξα μία ματιά γύρω-γύρω και είδα έναν βουλευτή, ο οποίο μπορεί να μην μίλησε καθόλου, αλλά μπορεί να γράφει ε, προτάσει συνέχεια. Μπορεί κάποιος άλλος ε, να μην έγραψε καμία πρόταση, καμία τροπολογία. Άλλοι βουλευτές από εκεί που δεν μίλησαν καθόλου, άλλοι βουλευτές ήταν παρόντες, έλαβαν το λόγο, κάποιοι άλλοι ήταν παρόντες εν μέρη, παρακολουθούσαν όμως ε, και πότε μπορεί να έγραφαν και καμιά τροπολογία και πότε μπορεί να παρακολουθούσαν τη συζήτηση λίγο και να μίλησαν. Κάποιο άλλο που ξέρω ήταν παρόν όλη την ώρα, είμαι σίγουρο ότι έγραφε τροπολογίε. Γιατί όποτε τον κοίταγα έβλεπα ότι κάτι παρακολουθούσε άσχετο με τη συνεδρίαση. Πώς θα μετρήσουμε λοιπόν ποιος είναι ο καλός βουλευτής και ποιος είναι ο λιγότερο καλός. Κάποιοι έχουν την εντύπωση ότι υπάρχει κάποιο μετρητής ε, βουλευτική δραστηριότητα που μπορούμε να πάρουμε μέσα σε μια συνεδρίαση επιτροπή και να μετρήσουμε τη δουλειά των βουλευτών. Δεν υπάρχει τρόπος να γίνει αυτό. για τα κτίρια και τα χρήματα που θα πρέπει να διαθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ναι, έχουμε πολύ συχνά κοινά κτίρια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις χώρες, αλλά δεν είναι πάντα τόσο αγαστή η συνεργασία. Πρέπει και αυτό να το, να το ε, αναφέρουμε. Και αντίστοιχα να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να προβούμε στα κατάλληλα ε, συμπεράσματα και τις συνέπειες. Πρέπει να το συστήσουμε λοιπόν. Και επίσης ηλεκτρικά οχήματα. Δεν υπάρχει επιλογή για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στο Στρασβούργο. Τόσο άλλως είναι αρκετά δύσκολο να βρούμε αυτοκίνητα στο Στρασβούργο. Αρκετά για όλους. Το αν θα πρέπει να τα μεταφέρουμε από εδώ εκεί, τι να σας πω. Άλλη επιλογή δεν υπάρχει. Είναι δύσκολο και το θέμα των ταξί. Χώρος στάθμευσης δεν υπάρχει. Να μην μιλήσω για το αεροδρόμιο. Αυτά. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για όλες αυτές τις διευκρινήσεις σας. Ευχαριστούμε και για τις προτάσεις που κάνετε. Όλοι, και οι μεν και οι δε, πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν όσον αφορά το κόστος του Κοινοβουλίου και όσον αφορά και την αποτελεσματικότητα του Κοινοβουλίου. Μιλάμε για προστιθέμενη αξία. Εμείς πρέπει να αποδείξουμε ότι υπάρχει αυτή η κοινοβουλευτική προστιθέμενη αξία αν η δημοκρατία δεν έχει τιμή, έχει όμως ένα κόστος. Και στους χρόνους που ζούμε, στους καιρούς που ζούμε, πρέπει να ελέγξουμε τις δημόσιες δαπάνες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Ήταν η πρώτη ανταλλαγή απόψεων που είχε η Επιτροπή μας για αυτό το θέμα. 9 Μαρτίου στις 12 είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Οι τροπολογίες θα συζητηθούν στις 7 Απριλίου όταν θα εγκρίνουμε και την τελική έκθεση, η οποία θα έρθει κατά πάσα πιθανότητα 13 Απριλίου στην Ολομέλεια προς ψήφιση. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που μας βοηθήσατε να ελέγξουμε τις δημόσιες δαπάνες και να βοηθήσετε την αρχή με προπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα τώρα το οποίο όμως δεν έχει δυσκολίες, είναι το ελεγκτικό συνέδριο που αντιμετωπίζει δυσκολίες επειδή δεν καταφέρνει να προσλάβει τους συνεργάτες που χρειάζεται. Προτείνει λοιπόν τρεις μόνιμες θέσεις, AST3 και μία θέση AST1, να τις κάνουμε τέσσερις ε, θέσεις AST3 προσωρινών υπαλλήλων. Κάτι το οποίο δεν δημιουργεί καμιά δυσκολία για μας. Ο συνάδελφος ο Δεπρέ μου ανέθεσε να σας πω ότι εκείνος συμφωνεί και άρα θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε κι εμείς και να ενθαρρύνουμε το ελεγχτικό συνέδριο να εφαρμόσει αυτά τα οποία επιθυμεί. Παρατηρήσεις, αντιρρήσεις, όχι. Καλώς. Εγκρίνεται λοιπόν. Εξαντλήσαμε εδώ την ημερήσια διάταξη. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να συζητήσουμε? Όχι από ό,τι βλέπω. Έλξη συνεδρίαση.